Αγαπητοί συνάδελφοι, κηρύσω την έναρξη της συνεδριάσεως εκφράζοντας τη χαρά μου ε, που έχουμε σήμερα προσκεκλημένο τον Υφυπουργό κύριο Καλέντα, Υφυπουργό Εμπορίου, που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου στα θέματα του Διεθνούς Εμπορίου έχουμε μια σειρά από σημαντικά θέματα που εκλήθη να διαπραγματευτεί η Προεδρία της Ιταλίας. Ιδιαίτερα για το TTIP και το ΚΕΤΑ, ΣΕΤΑ, τα πολύ σημαντικά αυτά θέματα. Αλλά επίσης και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με εμπορικές συμφωνίες. Τα δύο νομοθετήματα λοιπόν που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το TDI και το IPI θα μας εκθέσει επίσης καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η εμπορική πολιτική μπορεί να οδηγήσει επιστορές εργασίες και ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη. Καλώς ήρθατε. Η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε στο παρελθόν απεδείχθη πολύ συνεργατική. Εύχομαι και στο μέλλον η συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου να είναι το ίδιο καλή. Ευχαριστώ που ήρθατε λοιπόν και σας δίνω ευθύς αμέσως το λόγο. Χίλια ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε και μέλη της Επιτροπής. Τώρα προσεγγίζουμε ε, το τέλος ε, του εξαμήνου της Ιταλικής Προεδρίας και έχω την ευκαιρία να τοποθετηθώ εκ νέου ενώπιον αυτής της Επιτροπής για να αναφερθώ σε έναν απολογισμό στον τομέα της εμπορικής πολιτικής για το τελευταίο εξάμεινο. Θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στους νομοθετικούς φακέλους, καταρχήν για δύο σχέδια κανονισμού για τον εξεχρονισμό κανονισμό των ε, μέσων εμπορική Άμυνα ε, και για το μέσο για τι δημόσιε προμηθείες, για του δημόσιου διαγωνισμού, όπω ε, είναι γνωστό και ω μέσο βιβαιότητα. Η Ιταλική Προεδρία έχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά τα δύο θέματα για να καταλήξει σε συμβιβασμό στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό των μέσω εμπορική άμυνας, εν λόγω πρωτοβουλία εστάλει από την Κομισιόν ε, ήδη από το 2012, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα μηχανισμό για να μπορεί να ανταποκριθεί σε αθέμητες συμπεριφορές από τρίτες χώρες. Πέρα από να το αποκαταστήσει στους κανόνες για όλους, ε, σε σχέση με τις ε, χώρες που έχουν πολύ αποτελεσματικούς κανόνες TI επίσης για να έχουμε ένα μέσο για να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις μας από τον αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι στην ανάγκη να απαντήσουμε στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον κόσμο των επιχειρήσεων προσπαθήσαμε να ε, απευθυνθούμε στα κράτη-μέλη και να τα πείσουμε προκειμένου το Συμβούλιο να αναλάβει το ρόλο του συνομοθέτη για να απαντήσει ε, στο νομοθέτημα που παρουσίασε η Κομισιόν. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτού Αναμένω ότι σε αυτό το φάκελο υπάρχουν πολύ διαφορετικές ευαισθησίες εντός του Συμβουλίου. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βρούμε μια γραμμή συμβιβασμού ε, που να καλύπτει τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών. Παρόλες τις προσπάθειες που κάναμε για να προχωρήσει αυτός ο φάκελος και να κατορθώσουμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε το διάλογο με το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο δεν κατόρθωσε να ξεπεράσει τις εσωτερικές ε, διαφωνίες και στις 21 Νοεμβρίου δεν μπορέσαμε παρά να διαπιστώσουμε την κατάσταση αυτή και να ξεκινήσουμε ένα στάδιο εσωτερικού προβληματισμού όπου το κάθε κράτος μέλος ανάλογα ε, με το παραγωγικό του σύστημα να μπορέσει να φτάσει σε ένα σύνθεση των θέσεων σε ό,τι αφορά το International Procurement Instrument, ξεκινώντας από τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τροποποίησης που είχε υποστηρίξει και την πρόταση της Κομισιόν, η Ιταλική Προεδρία εδώ προώθησε μία ε, πρόταση συμβιβασμού στα κράτη-μέλη, όμως και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην προηγούμενη, παρά τις προσπαθίες μας, δεν έγινε καμία πρόοδο σε τεχνικό επίπεδο το τελικό αποτέλεσμα είναι δυστυχώς πολύ απογοητευτικό. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς εντός, εκτός μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν ε, δυστυχώς διακριτική μεταχείριση. Αλλά ενώ ο κανονισμό enforcement ήδη δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μέσο για να αντιμετωπίσει καταστάσει όπου χώρε με τι οποίε έχουμε συμφωνίε για τι δημόσιε συμβάσει, δεν σέβονται του κανόνε που έχουν συμφωνηθεί, δεν υπάρχει ακόμα ένα μέσο για να καταπολεμήσουμε ε, τις αθέμικες ε, πρακτικέ ε, των εταίρων που δεν έχουν συνάψει με εμά συμφωνία. Το τελευταίο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου, Ιταλική Προεδρία, δουλειά διαπίστωσε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν δυσκολίε και διαφωνίε μεταξύ των κρατών μελών και σε ορισμένε περιπτώσει, φαίνεται ε, να σέβονται περισσότερο τι εθνικέ απαιτήσει παρά να προσανατολίζονται προ ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι η πρόσβαση στους δημοσιογονισμού πρέπει να είναι ευρωπαϊκό φάκελο και η Προεδρία μας θα να μην διακοπεί η συζήτηση για αυτό το θέμα και το Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά θεωρεί ότι δεν υπάρχει απάντηση, όμως έχουμε καθήκον απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες να βρούμε εναλλακτική μέσω του κατάλληλου προβληματισμού στις τεχνικές ε, συνεδριάσεις και με τη βοήθεια της Κομισιόν. Όπως σας είπα στην τη συνεδρίαση ε, του επίσημου συμβουλίου στις 21, δυστυχώς και εντός του συμβουλίου, υπήρχαν θέσεις ε, που δείχνουν ότι υπάρχει ιδεολογική ρήξη. Και για το λόγο αυτό Ακόμη και το να οικοδομήσουμε μέσα άμυνας, όχι μόνο να τα χρησιμοποιήσουμε, για ένα μέρος των μελών του Συμβουλίου αποτελεί κάτι που φτάνει στον προδοξιονισμό η Ιταλική Προεδρία δεν θεωρεί ότι κάτι τέτοιο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Να έχουμε μέσα εμπορική άμυνα δεν σημαίνει ότι θα τα χρησιμοποιούμε και με μη κατάλληλο τρόπο. Κατά την ε, δεύτερο εξάμεινο του 2014, η Προεδρία πολλέ φορέ ξεκίνησε και μια συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών για την κατάσταση των εργασιών για τον ΠΟΕ, κυρίω ε, κατόπιν του τέλματο ε, από τον περασμένο Ιούνιο για την υιοθέτηση του πρωτοκόλου για τη διευκόλυνση του εμπορίου. Ευτυχώς τις τελευταίες εβδομάδες μετά από τις ειδικές εξελίξεις ε, για ε, το ΙΤΑ. Μπορέσαμε να σημειώσουμε ότι υπήρχε μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Κινδίας σε θέματα επιστηστικής ασφάλειας. Ε, στις 27 Νοεμβρίου το Συμβούλιο του ΠΟΕ ενέκρινε τρεις σχετικές αποφάσεις. Καταρχήν το πρωτόκολλο για την οθέτηση συνθήκης για διευκόλυνση των πορείων των facilitation για το θέμα της αποθεματοποίησης τροφίμων για επιστηστική ασφάλεια και τη δουλειά μετά τον Παλί που θα καθοριστεί με τον Ιούλιο του 2015. Πρόκειται για πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για τον ΠΟΕ και για το πολυμερές σύστημα που ξεπερνά το τέλμα που είχε δημιουργηθεί και δίνει συνέχεια μετά τον Μπαλί. Επίσης το Συμβούλιο θα ξεκινήσει εκ νέου τις εργασίες ε, για τον ΠΟΕ και για τις αποφάσεις για την υπουργική διάσκεψη και για τον καθορισμό ενός νέου συγκεκριμένου προγράμματος εργασίας ε, για να ολοκληρωθεί η υπόλοιπη διαδικασία με προσπάθειες της Προεδρίας μας αφιερώθηκαν σε μια διατηλαντική σχέση μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών εδώ. Όπως είχαμε πει και στην πρώτη ακρόση, μέσω ομόφωνης ψηφοφορίας Συμβουλίου κατορθήσαμε να, να δημοσιευτεί η εντολή στο διαδίκτυο και επίσης να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Όλο αυτό σημειώνει ένα πολύ μεγάλο βήμα στον τομέα της διαφάνειας ε, και ε, στη συμφωνία μεταξύ θεσμών και Ευρωπαίων πολιτών. Ε, πέρα από τη συγκεκριμένα αποτελέσματα και συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν για την TTIP από εμά θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και στους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και στους Αμερικανούς. Καταρχήν τη δέσμευση των κρατών μελών ε, στο Συμβούλιο να δώσουν μια όθηση για μια δυναμική, για να έχουμε μια φιλόδοξη και δυναμική συμφωνία για να υπάρχει απελευθέρωση ε, στις ανταλλαγές ε, και στις επενδύσεις για να ενισχύσουμε την απασχόληση και να υπάρχει οικονομική μεγέθυνση. Δεύτερον, να αυξήσουμε το επίπεδο της διαφάνειας. Υπάρχει μια νέα στρατηγική επικοινωνία από την Κομισιόν που θα συζητηθεί αύριο στην TPC. Στις αυτή, σε αυτή τη στρατηγική δεσμεύεται τα μάλα η Ιταλική Προεδρία για ε, το υπόλοιπο χρόνο της Προεδρίας, στρατηγική επικοινωνίας και διαλόγου ενάντια της κοινωνίας των πολιτών και της κοινή γνώμης, υπογραμμίζοντας ε, τα κυρία σημεία της συμφωνίας και τα ωφέλη για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, κυρίως για τις μικρές και μισές επιχειρήσεις. Και εδώ κάναμε μια προσπάθεια σύνθεσης για να μπορέσουμε να ε, δεχτούμε τις διάφορες προτάσεις των αντιπροσωπιών Φυσικά προσπαθώντας ε, να έχουμε ξεχωριστά συμπεράσματα για την τίτυπα από τα συμπεράσματα για το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ο στόχος ήταν να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους Αμερικανούς χαράκτες πολιτικές, πολιτικής ε, ε, γιατί είχαμε κάποιες εξελίξεις και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ό,τι αφορά τώρα την ουσία στρατηγική της Ιταλικής Προεδρίας για την εμπορική πολιτική ε, καθόλου το εξάμεινο είχε ως προτεραιότητα να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε έτσι ώστε να μπορούν να ολοκληρωθούν το αργότερο στα τέλη 2015 αρχές 2016 εκμεταλλευόμενοι το παράθυρο ευκαιρίας ε, που υπάρχει τώρα ε, μέχρι την έντονη προεκλογική διαδικασία ε, για τις προεδρικές εκλογές. Ε, χρειάζεται πολύ φαντασία για να ε, κατανοήσουμε ότι το 2017 αν δεν ολοκληρωθούν διαδικασίες θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθεί σε μια τελείως διαφορετική διαπραγματευτική θέση ενώπιον των ΗΠΑ καθώς οι Ηνωμένε Πολιτείες αναπτύσσονται νότερα από εμά και η TPP θα έχει ολοκληρωθεί ήδη για εδώ και δύο χρόνια. Με την κυρία, η κυρία Μάστρομ θα, συζητηθεί με τον, θα συναντηθεί με τον κύριο Φρόνμαν προκειμένου να μπορέσουν να βρουν τις landing zones μεταξύ φιλοδοξίας και ρεαλισμού σε ό,τι αφορά το STS που σε λίγες εβδομάδες θα μπορούσε επίσης να συζητηθεί για τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που ξεκίνησε από την Κομισιόν τους προηγούμενους μήνες θα θέλω να σας πω και πριν να ξεκινήσει οποιαδήποτε πρωτοβουλία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να σκεφτεί το θέμα αυτό προσεκτικά, αν χρειάζεται στο να προχωρήσουμε σε συζήτηση και σε μία ε, ρητή αίτηση να εξαλειφθεί ο μηχανισμός αυτός ε, εντός ε, των διαπραγματεύσεων TTIP. Πρέπει να ξέρουμε πόσο σοβαρές συστημικές συνέπειες θα έχουμε για το μέλλον, όλη, για όλο το μέλλον της πολιτικής επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ένα αποτέλεσμα ντόμινο βάσει και όσων έχουμε διαπραγματευτεί με τον Καναδά και με τη Σιγκαπούρη και θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα και στο μέλλον στις διαπραγματεύσεις μας με την Κίνα επίσης ε, θα μπορούσαν να υπάρχουν αντίπεινα ε, παραδείγματο χάρη σε τομείς που σε ενδιαφέρουν όπως οι διαγωνισμοί και κατόπιν υπό το φως της συνθήκης της Αβώνας θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει το μηχανισμό DSDS ε, διατηρώντας ε, ε, σε αντίθετη περίπτωση πάρα πολλές ξεχωριστές διμερείς συμφωνίες. Δεν μπορώ να σκεφτώ το Κοινοβούλιο θα ταχθεί η συνθήκη της Λαβώνας και θέλω να σας διαβάσω κάτι που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σχετικό το συμπέρασμα των ε, συνθήκων, ε, των διμερών συνθήκων, ε, κυρίως με τις μεταβατικές χώρες, δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο για άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό. και συνθήκη αυτή θέτει την νομική θέση για τους επενδυτές, όπως τον έχουν ίση μεταχείριση, απαγορεύει μέτρα διάκρισης, προβλέπει ίση μεταχείριση με τη χώρα ή με την εθνική εταιρεία πρόσθετα. Γενικά δίνουν στους επενδυτές την επιλογή να σκίσουν τα δικαιώματα αυτά, δική τους πρωτοβουλία ε, προσφεύγοντας σε ουδέτερα διεθνή δικαστήρια έτσι λοιπόν αποφεύγοντας ε, να έχουν απρόβλεπτους παράγοντες αν προσφυγούν στα εθνικά δικαστήρια ακόμη και με την, ε, μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας οι διμερεί συνθήκες που ισχύουν τώρα με πάνω από 130 χώρες αποτελούν μία βάση για να υπάρχουν επενδυτικές εγγύσεις. Αυτό προέρχεται από γερμανική έκθεση για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ε, Ενώ καταλαβαίνετε ότι ε, το να κάνουμε ως θέμα της διμερής πολιτικής ε, της αυτές τις διμερείς συμφωνίες ε, να τις θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητα και να λέμε ότι από την άλλη δεν μπορεί να το αγγίξει αυτό η Ευρώπη είναι κάπως αμφίσιμο. Επίσης, το Νοέμβριο υιοθετήθηκαν γενικά συμπεράσματα που είχαν προταθεί από την Ιταλική Προεδρία τις προηγούμενες εβδομάδες και ε, έγιναν κάποιες προσπάθειες ε, από όλα τα κράτη-μέλη για τη διατύπωση. Τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν ότι η στρατηγική για το εμπόριο είναι ουσιαστικό τμήμα της πολιτικής για την ανάπτυξη και επομένως πρέπει να συνάδουμε τις άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συμπεράσματα βασίζονται κυρίως σε όσα ε, είπε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο και στην εξωτερική διάσταση του εμπορίου ως απαραίτητο μέσο για να ευνοηθεί η εμπορική μεγέθυνση και απασχόληση. Με αυτό το έγγραφο το Συμβούλιο καλεί ε, τον Επίτροπο Εμπορίου να ξεκινήσει μια διαδικασία για την επικαιροποίηση της στρατηγικής για την εμπορική πολιτική υπό το φως του νέου οικονομικού πλαισίου και σύμφωνα ε, με τα κριτήρια της Επιτροπής. Και εμείς ευχόμαστε εντός όλου αυτού του προβληματισμού να κλείσει αυτό το λογικό ρήγμα εντός ε, του Συμβουλίου για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια συμφωνία στο νομοθετικό επίπεδο. Κατά την Προεδρία μας ε, κάναμε σημαντικά βήματα προς τα μπρος και στις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών με την Ιαπωνία Καταρχήν ολοκληρώθηκε η ετήσια αναθεώρηση της ρήτρα ραντεβού για τις διαπραγματεύσεις με το Τόκιο υπό το φως της καλής θέλησης που έδειξε η Ιαπωνία για να υπάρξει άρση των μη δεσμολογικών εμποδίων βάση του οδικού χάρτη που είχε καταρτιστεί δεύτερον τον Οκτώβριο ε, μπορέσαμε να προχωρήσουμε στην ε, ε από τον καταλογιά της ε, τρεις ε, εταιρείε σιδηροδρομικέ ε, στην Ιαπωνία και είχαμε και τον 7ο γύρο διαπραγματεύσεων με την Ιαπωνία και μπόρεσε να δοθεί νέα όθηση στις διαπραγματεύσεις με ένα τόσο σημαντικό οικονομικό εταίρο και στρατηγικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να αναφορώ και στη Συμφωνία Ελεύθερων Συνολογών με το Βιετνάμ. Είναι πιο προηγμένε οι διαπραγματεύσει και ίσω θα μπορούσε να συναυθεί συμφωνία στην άνοιξη του 2015. Πάντω παραμένουν κάποια λεπτά θύματα όπως η προστασία γεωγραφική ένδειξη, θέματα που έχουν να κάνουν με τις κρατικές επιχειρήσεις που πρέπει να συζητηθούν στο τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων και το Συμβούλιο θα συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή. Πάντοτε σε ό,τι αφορά τη χορήγηση αυτόνομων προτιμήσεων, η Προεδρία κατόρθωσε να λάβει την έγκριση του Συμβουλίου και ε, με την υιοθέτηση χωρίς τροπολογία στην Επιτροπή τα, ε, ότι θα υπάρχουν νέες ε, αυτόνομες προτιμήσεις για τη Μολδαβία και επίσης η Ιταλική Προεδρία είχε δεσμευτεί για να προχωρήσει για άλλα δύο θέματα που ενδιαφέρουν πολύ την εμπορική πολιτική για τα Δυτικά Βαλκάνια καταρχήν, η Κομισιόν προτείνει να υπάρχουν η μεγαλύτερη διάρκεια των προτιμησιακών μέτρων για τις χώρες που αποτελούν τμήμα της πρώην Ιουκοσλαβίας το κανονισμό 1215 του 2009. Τώρα για το 2020 υπάρχουν κάποιες Υποθέσει για το Εκουαδόρ από το 2014 τον Ιούλιο ολοκληρώθηκαν συναλλαγές, οι διαπραγματεύσει για τη Συμφωνία Συναλλαγών και με την Κολομβία και το Περού. Η Κομισιόν εθέτησε την πρόταση κανονισμού COM 2014-585 ε, και προκειμένου να αποφύγουμε ότι με την έξοδο του Εκουαδόρ να υπάρξουν δασμοί που θα εισαχθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κανονισμός αν δεν θετηθεί, θα έχει συνέπειες τελωνιακές και εμπορικές και θα σήμαινε πολύ μεγάλη ζημία ε, για τους οικονομικούς φορείς. Έτσι λοιπόν πρέπει να υιοθετηθεί γρήγορα αυτός ο κανονισμός ε, και έχουν προταθεί και κάποιες τροπολογίες από την ίντα όπως στην περίπτωση ότι αν υπάρχει παραβίαση των πολιτικών ρητρών η απόφαση για την αναστολή των προτιμήσεων πρέπει να λάβει τη μορφή κατεξουσιοδότηση πράξεων αντί εκτελεστικής πράξης, όπως προτείνεται από την Κομισιόν με τη συνένεση του Συμβουλίου και με την έγκριση της νομικής υπηρεσίας του. Τέλος, κατά τη διάρκεια του εξάμεινου της Προεδρίας, η Κομισιόν ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες ε, με τρεις ε, περιφέρειες, τη Δυτική Αφρική, την ε, κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής και την κοινότητα για την Νότια Αφρική. Πρόκειται για τρία σημαντικά θέματα γιατί θα υπάρχει διευκόλυνση στην αγορά για τους μικρούς γεωργούς των περικλειστών ζωνών. Επίσης, σε χάρη στην ολοκλήρωση αυτών των συμφωνιών, οι χώρε χώρες θα συνεχίσουν να έχουν προτιμησιακή μεταχείριση ε, προκειμένου να έχουν πρόσβαση τα εμπορεύματά του στι αγορέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έχουμε και το νέο Market Access Regulation στην Δυτική Αφρική. Η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί πριν από το τέλο τη Ιταλικής προεδρία. Σα ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την περιεκτική παρουσίασή σας. Και νομίζω κατέστη πλέον σαφές ε, ότι πραγματικά ένα ιδιαίτερα ενεργό ρόλο έχετε ως ε, προεδρεύουσα ε, χώρα του Συμβουλίου ώστε να προαχθούν αυτά τα θέματα. Θέλω ιδιαίτερα τις προσπάθειές σας να τις αναγνωρίσω και να τις τονίσω για την επίτευξη κάποιας λύσης στο Συμβούλιο και θα το έλεγα και εντελώς ξεκάθαρα και θα το τόνιζα αυτό που είπατε. Δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου το ότι ένα από τα κράτη-μέλη αυτό το μέσο εμπορικής άμυνας το οποίο σε μια περίοδο παγκοσμιοποιημένου εμπορίου είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείται το παρακολεί μέσω δηλαδή εμπορικής αμυντικής ε, ε, πολιτικής ε, και έχουμε πολλές συμφωνίες ε, εμπορίου και δεδομένου αυτού του στοιχείου είναι τεράστια σημασία να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο πλαίσιο δικαίου ώστε να μπορούμε να έχουμε τέτοια μέσα προστασίας ε, των εμπορικών μας συμφερόντων. Μπορώ να σας υποστηρίξω λοιπόν να γίνει ό,τι περνάει από το χέρι σας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να είναι μια στεναρή εντολή προς το Συμβούλιο ώστε να μπορέσουμε άμεσα να περάσουμε στις διαπραγματεύσεις και εμείς από το Κοινοβούλιο είμαστε πρόθυμοι πραγματικά ταχύτατα να εξεύρουμε ένα συμβιβασμό, να αναζητήσουμε για να εξεύρουμε ένα συμβιβασμό για την σωστή χρήση αυτού του σύγχρονου μέσου εμπορικά. Μην χαλαρώσετε λοιπόν στο Συμβούλιο και να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια να πείσετε τα κράτη-μέλη. Σε ένα πρώτο γύρο θα λάβουν τον λόγο να παρέμουν οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων. Μετά θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο με ευρωβουλευτές. Από το ο κύριος Κασπάρη δεν παρίσταται. Ποιος θα λάβει τον λόγο. Ο κύριος Κέλλη ζήτησε τον λόγο για το ΕΛΚ. Παρακαλώ κύριε Κέλλη. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πράγματι για μια πολύ περιεκτική πλήρη επισκόπηση για τις ε, τη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων. Η λειτουργία αυτή υπό κάποιες πτυχές ε, που λειτουργήσε καλά ήταν ένας ιδιαίτερα στρατηγικός ρόλος της ε, Προεδρίας. Λαμβάνοντας υπόψη ε, την προηγούμενη προσπάθεια στην προηγούμενη θητεία για να μπορέσουμε να κινηθούμε προς τα εμπρός, να σημειωθεί πρόοδος, είδαμε όλη την δημιουργία της νέας Επιτροπής που συγκροτήθηκε και το τι γίνεται πίσω από τα σκηνικά θα πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθούν αυτές οι προσπάθειες ιδιαίτερα να γίνει η πρόοδος για τις συμφωνίες που ήταν σημαντική πρόοδος που επετεύχθη στις εμπορικές ε, συμφωνίες με πολύ συνετό και λογικό τρόπο η πρόοδος αυτή που σημειώθηκε σε όλες τις γενικές συζητήσεις. Ένα σημείο θέλω μόνο να ερωτήσω και είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό που ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει να αποσαφινιστούν τα πράγματα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Οι σχέσεις με το ISDS, ιδιαίτερα όσον αφορά την TTIP, τη Συμφωνία Επενδύσεων και Εμπορίου με τις ΗΠΑ. Και σε σχέση με το όπως το βλέπουν πολλοί ότι είναι κάτι κακό λέει και επικίνδυνο και που θα το χρησιμοποιήσουν και θα το εκμεταλλευτούν επιχειρήσεις αποκλειστικά προς όφελός τους. Ίσως εδώ υπάρχει κάποια έλλειψη γνώσης γεγονότων. Ίσως η ε, Ιταλική Προεδρία θα μπορούσε να διοργανώσει μια κρόαση στο επίπεδο της δικής μας ε, Επιτροπής για να γίνει κατανοητό, κατανοητό τι συμβαίνει, πόσες φορές ε, έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες χρήσης αυτών των μέσων ώστε να έχουμε μια επίσημη πλέον θετική, ε, θετικά διαρθρωμένη συζήτηση με πραγματικά αντικειμενικά στοιχεία γνώσης ε, για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση με αυτές τις προκλήσεις. Νομίζω θα ήταν πολύ θετικό αυτό για την Ιταλική Προεδρία να στέψει με επιτυχία την Προεδρία της ε, μια τέτοια εκδήλωση. Ευχαριστώ. Για τους ε, σοσιαλδημοκράτες η Αλέσια, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε για αυτή την πολύ λεπτομερή παρουσίαση του έργου της Προεδρίας. Εγώ θέλω να κάνω τρεις γενικές παρατηρήσεις, γιατί οι συνάδελφοι θα μπουν ε, περισσότερες λεπτομέρειες των μονομένων θεμάτων. Καταρχήν, θέλω να ξεκινήσω από ένα θέμα ουσίας σε ό,τι αφορά την εμπορική πολιτική, δηλαδή το θέμα του πώς μπορούμε να επιτεχύνουμε τη θέση σε των εμπορικών συμφωνιών, γιατί ακόμη και χτες τη συζήτηση που είχαμε με την Επιτροπό διεφάνει από όλες τις πολιτικές ομάδες η αναγκαιότητα να μπορούμε να έχουμε το συντομότερο δυνατόν σε ισχύ συμφωνίες που ε, χρειάζονται κατά καταναλώνουν πολύ χρόνο. Δηλαδή από τη συμφωνία να μπούμε στη θέση σε ισχύ μετά από δύο ή τρία έτη στην καλύτερη περίπτωση είναι φυσικά ένα πρόβλημα δεδομένης ε, τη ταχύτητα με τις οποίες κινεί το κόσμος. Οι άλλες χώρες λαμβάνουν αποφάσεις και δεδομένης και της αναγκαιότητας να δώσουμε και στις δικές μας επιχειρήσεις μια βεβαιότητα σε σχέση με τις ευκαιρίες που έχουν. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία για την ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με τη διαφάνεια. Εκτιμήσαμε πολύ την προσπάθεια που έγινε από την Ιταλική Προεδρία καταρχήν ε, οδήγησε σε απεμπλοκή με τη δημοσιοποίηση της εντολής και με την ε, νέα στρατηγική που παρουσιάστηκε την εβδομάδα την Κομισιόν. Εδώ θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει ένα ακόμη βήμα προς τα μπρος, δηλαδή πώς ε, από αυτή τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, των διαπραγματεύσεων, να μπορούμε να φτάσουμε σε πραγματική διαφάνεια που φυσικά αυτό αφορά και το Κοινοβούλιο με τον προδραστικό ρόλο που πρέπει να έχει σε σχέση με τους πολίτες, αλλά και το Σύμφωνο και αυτό, όχι μόνο για τη διατηλαντική εταιρική σχέση λόγουν και επενδύσεων, αλλά και για τις άλλες εμπορικές συμφωνίες. Πρέπει να καταλάβουμε πώς και το Συμβούλιο μπορεί μαζί με το Κοινοβούλιο να προωθήσει δράσεις συμμετοχής των πολιτών. Και τελευταία σκέψη. Και είναι μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Ποιες πιστεύετε μπορείτε να είναι οι προτεραιότητες ε, για, ε, που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην νέα ανακοίνωση. Η Επίτροπος ε, χτες μας ανακοίνωσε ότι τις επόμενους μήνες θα παρουσιαστεί αυτή η ανακοίνωση. Επομένως, ποιες πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οι προτεραιότητες που θα ενταχθούν σε αυτή την ανακοίνωση που θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Εμπορικής Πολιτικής. Ευχαριστώ. kein Mandat. Dann, äh, Η Μαρίκε τώρα, παρακαλώ. Thank you. Chair, thank you, Minister. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ. Για την παρουσία σας ακούσαμε αρκετά για την TTIP. Ήταν μάλλον ασαφή βέβαια αυτά που μας είπατε για την TTIP. και βλέπω ότι δεν ε, υπάρχει δεν υπάρχει πρόθεση από το Συμβούλιο να συμμετάσχει. στις διαπραγματεύσεις. Είναι κάτι όμως το οποίο δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε. Χρειάζεται με τις ε, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να κοιτάξουμε τις διάφορες περιοχές, να κοιτάξουμε τους διάφορους τομείς και να αντιμετωπίσουμε θέματα τοπικά και εθνικά ενδεχομένως. Χαίρομαι που είναι δημόσια διαθέσιμη διαπραγματευτική εντολή. Απ' την άλλη όμως πήρε πολύ καιρό και πρέπει να μας απασχολεί στο ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος. Χρειάζεται η διαφάνεια, χρειάζεται όμως και η προσβασιμότητα στην πληροφορία και η βελτίωση της υποστήριξης των έργων. Έχετε κάποια συγκεκριμένη λοιπόν πρόθεση για το για την επιτυχία του μέσα από το Συμβούλιο, τι μπορείτε να κάνετε για να πείσετε περισσότερο τα κράτη-μέλη ότι είναι κάτι το πολύ σοβαρό και ότι χρειάζεται να βοηθήσουν και εκείνα για να προωθηθεί το θέμα αυτό. Να έχουμε περισσότερη ενημέρωση. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο που θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Αλλά πρέπει κάποια σημεία να τύχουν της απαραίτητης προσοχής. Και ορισμένα από αυτά δεν έχουν καμία προσοχή. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε τι μπορεί να γίνει. Και επίσης από τα τελευταία ε, τις τελευταίες εργασίες του Συμβουλίου έχουμε το θέμα της ε, διτής χρήσεως, στρατιωτικής και μη στρατιωτικής χρήσεως. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει τον τόνο και να ενσωματώσει και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συνεπειών σε αυτά από τις εξαγωγές ε, που είναι τελείως αρρύθμιστες των εξαγωγών τέτοιου είδους, τις εξαγωγές λοιπόν τέτοιου είδους υλικών και προϊόντων. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τεθεί στην πρωτοπορία. Ερωτώ λοιπόν το θέμα αυτό στον, σε επίπεδο Συμβουλίου πώς βλέπετε να προχωρεί. Γιατί το Κοινοβούλιο έχει δώσει όθηση, έχει πιέσει και την Επιτροπή, αλλά θα πρέπει και το Συμβούλιο να κινηθεί. Ευχαριστώ, η ευχαριστώ την Γκουε, μάλλον για για τους πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα επανέλθω στα σχόλια του Μπέρντ Λάγκε για τα μέσα βιομηχανικής άμυνας. Αφήνουμε ακόμα την πρωτοπορία στους Κινέζους για, τις για τα ε, φωτοβολταϊκά, πράγμα που καταστρέφει πολλές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και δεί στην Ιταλία. Πρέπει η Ευρώπη πλέον να βρει τον τρόπο να προστατευθεί. Επίσης, αναφερθήκατε στις ε, δημόσιες προμήθειες και την ε, αμοιβαιότητα. Συμφωνώ με την αμοιβαιότητα. Αλλά εάν η αμοιβαιότητα πρόκειται να θεσπιστεί με αρχή την Ευρω... της ευρωπαϊκής αγοράς, άνοιγμα δηλαδή των αγορών, με βάση τι αρχέ τη ευρωπαϊκή αγορά που συνεπάγονται απόλυτο άνοιγμα των αγορών, αντίθετα από αυτό που συμβαίνει στην διεθνή αγορά, γιατί ναι, μεν πρέπει παντού οι δημόσιες αγορές, ε, οι κρατικές αγορές να ανοίξουν και να γίνουν όπως στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και κάποια άλλα μέρη του κόσμου να αποτελέσουν ένα εργαλείο στρατηγικών επιλογών κτλ. Αλλά το άνοιγμα τώρα των αγορών θα ήταν τεράστιο σφάλμα. Για το TTIP. Τελευταία φορά που θα έρθει κύριε Υπουργέ, μας εξηγήσατε ότι οι θέση της Ιταλικής Προεδρίας ήταν η επιδίωξη μιας νέας εντολής πιο περιορισμένες αναδιαμορφωμένης με μια νέα στρατηγική. Και από την άλλη βλέπουμε με την έκθεση του Συμβουλίου του Νοεμβρίου ότι δεν αλλάζει τίποτα, τουλάχιστον από, την ανακοι... από το ανακοινωθέν ως προς την ευρωατλαντική αυτή συνθήκη. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς αξιολογείτε την πορεία όλη αυτή και τις δυσκολίε που αντιμετωπίσατε για να ξαναδιαμορφώσετε και να ε, βάλετε σε νέες διαστάσεις αυτή τη συνθήκη. ISDS. Η κατάσταση στην Ευρώπη σε κάθε επίπεδο δεν είναι και τόσο λαμπρή σε διπλωματικό, εμπορικό και άλλο επίπεδο. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε καταφέρει όλα τέλεια και δεν χρειάζεται να διορθώσουμε τίποτα. Ίσως θα έπρεπε να ξανά εισαγάγει ρυθμίσεις, άλλωστε το έχει παραδεχτεί αυτό για τα χρηματοπιστωτικά η Ευρώπη για το ISDS ε πρέπει να δούμε ότι δεν είναι απλώς ένα μέσο επικοινωνιακό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ε, Γερμανίας έχουν επανειλημμένως εκφράσει, όπως και άλλα, ε, όπως και εθνικά κοινοβούλια, παραδείγματι, την απόρριψή τους για το σύστημα ESDS. Γιατί λοιπόν η προστασία των επενδύσεων να, ερμηνε... να περνάει αναγκαστικά μέσα από έναν μόνο μηχανισμό που είναι αυτή η εξοδικαστική διευθέτηση των διαφορών, του ESDS. Βεβαίως είναι πολύ σοβαρές ε, οι ανησυχίες και τα μελήματα για την εθνική κυριαρχία των κρατών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο επικοινωνιακό, δεν είναι ότι δεν εξηγούμε καλά τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν οφείλεται σε αυτό το ότι ο κόσμος είναι εναντίον. Ε, ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος και έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω από το ΕΛΚ. Καταρχήν, σας ευχαριστώ όλους που είπατε ότι ήταν πολύ λεπτομερής η παρουσίασή μου. Ελπίζω να μην ε, πλήξατε. Πέραν αυτού. Για το θέμα το SDS, επίλυση διαφορών κράτους επενδυτή, ίσως θα πρέπει να δούμε κάποια θέματα που πάνε μαζί. Καταρχήν, ναι, πρέπει να οργανώσουμε μία συνάντηση μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν, ε, ίσως πάνω από μία συναντήση για αυτό το θέμα, επίλυση διαφορών επενδυτή κράτου και θα πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για αυτό το θέμα. Γιατί βλέπετε καταρχήν ε, ε, πρέπει να επιλεχθεί σωστά η εντολή διαπραγματευτική και λέει στη διαπραγματευτική εντολή ότι καμία ρήτρα του STS δεν πρέπει να προκρίνει ε, να ε, αντιτίθεται στη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των κρατών μελών να ασκήσουν την κυριαρχία τους. Και τώρα εδώ, αυτό που λέω και σας απαντώ είναι το εξής σήμερα Έχουμε ένα θέμα ότι χρησιμοποιείται το SDS ε, από τα ευρωπαϊκά κράτη και μάλιστα το ένα κατά του άλλου. Ε, στρέφεται κατά του άλλου και στις, ε, στο 50% των περιπτώσεων χρησιμοποιήθηκε από τους επενδυτές προς άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Τι πρέπει να κάνει το ευρωπαϊκό SDS. Πρέπει να είναι πολύ πιο περιορισμένο από αυτό που έχουμε στις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες και σύμφωνα με τη γνώμη της Προεδρίας θα πρέπει να απαντά σε δύο περιπτώσεις. Όταν ε, έχουμε μία απαλωτρίωση και όταν δεν υπάρχει αποζημίωση και όταν υπάρχει κατάφορη διάκριση. Αυτές είναι οι δύο περιπτώσεις για τις οποίες γεννάται το STS και δεν θα πρέπει να χειρογωγηθεί με άλλο τρόπο. Εγώ διάβασα πριν τη γερμανική έκθεση γιατί δεν θέλω σε αυτό το ζήτημα, το STS, γύρω από αυτό να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ε, και τελικά να καταλήξουμε ώστε να μείνουμε με τα εθνικά SDS που είναι πιο περιοριστικά και επικίνδυνα και μην αντιμετωπίσουμε το θέμα διαρθρωτικά και έξυπνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό να κάνουμε. Τώρα, για ε, το Μόσκο, τώρα έχουμε μία παράδοξη κατάσταση, γιατί θα ε, μεταφραστεί η συμφωνία σε 24 γλώσσες, έχει μονογραφηθεί. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι παράδοξο. Εγώ εκπροσωπώ μία από τις 24 γλώσσες, αλλά πιστεύω ότι στην περίπτωση αυτή το γεγονό ότι η Ευρώπη πρέπει να περάσει, να ξοδέψει 7-8 μήνες για τις μεταφράσεις ε, είναι πραγματικά κρίμα γιατί χάνουμε δυνατότητα ε, να οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μας ε, να προβούν σε εξαγωγές η επόμενη Προεδρία θα πρέπει να θέσει το θέμα αυτό ό,τι αφορά τώρα τη μετάφραση, δηλαδή τη νομική μετάφραση ε, των διεθνών συμφωνιών ε, να γίνεται η μετάφραση μόνο στα αγγλικά. Διαφάνεια για το πακέτο Μάλστρομ. Χτες ε, νομίζω ήρθε εδώ η Επίτροπος και είναι ισορροπημένη αυτή η δεσμή μέτρων. Εγώ πιστεύω θα την υποστηρίξουμε και ήδη στην TPC αύριο. Έδωσε στην ε, Επίτροπο όλη την υποστήριξη του Συμβουλίου, είτε στην TTIP να υπάρχει μια μεγαλύτερη μια δομή μεγαλύτερη διαφάνεια, είτε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώ αυτή η διαδικασία τη διαφάνεια μπορεί να καλύψει και άλλε διεθνεί συνθήκε, να γίνει δηλαδή ένα πρότυπο διαφάνεια. Ποιε είναι οι προτεραιότητε. Σήμερα σας λέω την γνώμη μου. Σήμερα βλέπουμε ένα μεγάλο παιχνίδι για τις εμπορικές σχέσεις. Και πιστεύω, αν εσείς ε, δείτε την έκθεση κομισιών για την αύξηση των ε, μη δεσμολογικών εμποδίων που έχουν φτάσει ε, στο 90% μέσα σε λίγα χρόνια, θα δείτε στις έξι πρώτες θέσεις είναι όλες οι χώρες BRICS. Τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι εμείς στις χώρες αυτές επιτρέψαμε να αναπτυχθούν έχοντας μια ανισορροπία προστασίας και τώρα που έχουν μεσαία τάξη καταναλωτική προστατεύονται μέσω ε, ενός εργαλείου που εμείς δεν μπορούμε να επιτρέψουμε και είναι αυτά τα δασμολογικά εμπόδια. Δηλαδή, για μας ε, δεν έχει φτάσει ακόμη κάτι τέτοιο και κάτι τέτοιο δεν ε, μπορεί ε, να χρησιμοποιηθεί σε κρυφές διαδικασίες. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό εγώ νομίζω ότι τώρα πρέπει να κλείσουμε και να συμφωνήσουμε για την τύπη και για τις άλλες συμφωνίες με τις οποίες διαπραγματευόμαστε. Αν εσείς βάλετε μαζί όλο αυτό το, όλη αυτή τη ζώνη, θα φτάσουμε στο 63% του παγκόσμιου ΕΧΠ. Είναι ένας μεγάλος χώρος ελεύθερων συναλλαγών. Πρόκειται για χώρες που έχουν δεχτεί να παίξουν ισορροπημένα για την παγκοσμιοποίηση. Και αυτό πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να ασκήσουμε πίεση στις άλλες χώρες, στις BRICS και στις άλλες, που δεν συμφωνούν ε, έτσι ώστε στο δεύτερο στάδιο της ε, παγκοσμιοποίησης να αποφύγουμε κάτι που στο πρώτο στάδιο προκάλεσε προβλήματα στη Δύση. Εγώ νομίζω αυτή είναι η απόλυτη προτεραιότητα και αν ε, εμείς τώρα αρχίζουμε να εγκαταλείπουμε κάποια ρητορική που ίσως έχει κουράσει για τον πολυμερισμό και τα λοιπά και αρχίσουμε να δίνουμε μεγαλύτερη ε, σημασία στο εθνικό συμφέρον τη Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτό θα συμβάλλει και στον ελευθερό ανταγωνισμό. Τώρα για την διαφάνεια, για την... Εγώ συμφωνώ για το συμπέρασμα σας, γιατί το είπα, Νομίζω ότι το συμπέρασμα δήλωσε ξεκάθαρα ότι πρέπει να επιταχύνουμε, να συνάψουμε το συντομότερο τη συμφωνία και να μείνουμε στην εντολή. Ποτέ δεν ανέφερα το γεγονό ότι θα άλλαζα την εντολή. Σε αυτό το στάδιο να αλλάξουμε την εντολή σημαίνει ότι κλείνουμε τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες και φυσικά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου μεγεθύνονται οι γεωπολιτικές απειλές, το ίδιο ισχύει για τις εμπορικές απειλές, όπως ανέφερα για ε, τα μετασμολογικά εμπόδια, πρέπει να έχουμε περισσότερη πρόσβαση στην αγορά και σύντομα πρέπει να το κάνουμε αυτό για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις μας. Ναι, ίσως το συμπέρασμα να έπρεπε να ήταν πιο ισχυρό. Αυτό ήταν το επίπεδο συνένεσης, το οποίο φτάσαμε και φυσικά λάβαμε τις υπόψεις και τις ευαισθησίες, αλλά... Το σημαντικό είναι ότι ξεκάθαρα από το Συμβούλιο πρέπει να κάνουμε αυτό σύντομα και εντός του πεδίου της εντολής. Δεν θεωρείται και δεδομένο. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για τη διαφάνεια. Φυσικά θέλουμε να δεσμευτούμε σε αυτό και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι καθήκον του κράτους μέλους. Πάντοτε αυτό το συζητώ και στο Κοινοβούλιο και με ΜΚΟ, με συνδικάτα, με όποιον θέλει να συζητήσει στην Ιταλία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και πρέπει να πω ότι μερικέ φορέ αντιπογοητεύομαι από το ότι όλοι ζητούν περισσότερη διαφάνεια και δεν διαβάζει την εντολή. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε να συζητούμε τις δημόσιες υπηρεσίες που δεν είναι συζήτηση, τις μειονικά οργανισμούς που δεν είναι στη συζήτηση για τη συνθήκη, την πολιτιστική εξαίρεση, τα οπτικοακουστικά. Όταν ε, λοιπόν ε, θα έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια πρέπει να την εκμεταλλευτούμε κιόλα. Τέλος. Για τις δημόσιες συμβάσεις και για τα φωτοβολταϊκά. Συμφωνώ μαζί σας. Όπως ξέρετε η Ιταλία ήταν πολύ, ε, ε πολύ έντονα ζήτησε μέτρα ε, έναντι της αθέμητης συμπεριφοράς της Κίνας. Και επίσης ε, είχαμε και κάποια αντίπεινα. Γιατί είναι σαφές, με συγχωρείτε, θα μιλήσω Ιταλικά. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και το πρόβλημα είναι ιδεολογικού χαρακτήρα. Το Μισό Συμβουλίο θεωρεί ότι οποιαδήποτε μορφή απάντησης, ακόμη και σε αφέμητες συμπεριφορές, είναι πρωτοξιονισμός και είναι ε, τεράστιο λάθος ε, γίνεται και για τα μέσα εμπορικής άμυνας και για τα φωτοβολταϊκά και για τις ε, δημόσιε συμβάσει. Αλλά αυτό πρέπει να το συζητήσουμε γιατί τι συμβαίνει και στο Κοινοβούλιο οι ίδιε χώρε που κατόπιν θέτουν βέτο στο Συμβούλιο κινδυνεύουν ε, να μπλοκάρουν οποιοδήποτε μέτρο. Α κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των δύο οργάνων γι' αυτό. Συγγνώμη για τις δημόσιες συμβάσεις. Ε, δεν μπορούμε να κλείσουμε την Ευρώπη ε, στις ε, ξένες συμβάσεις. δηλαδή τι τις χώρες που έχουν ανοίξει για μας. Γιατί όλες οι μεγάλες εταιρείες μας δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Με συγχωρείτε, ήταν πάρα πολλά τα θέματα που τέθηκαν και ίσως μίλησα πολύ. Ευχαριστώ. Και ένα γρήγορο δεύτερο γύρο ζητώντας συγγνώμη ε, από την EFDD γιατί σας λησμόνησα στον πρώτο γύρο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ παρακολούθησα πολύ προσεκτικά το έργο της Ιταλικής Προεδρίας αυτούς τους μήνες και μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών η Προεδρία είχε μια μεγάλη ευκαιρία για να καθορίσει τη στρατηγική και εγώ νομίζω ότι τελικά την έχασε αυτή την ευκαιρία, δεν την ανέπτυξε πλήρως. Αυτό ισχύει για το μέσο εμπορική Άμυνα, που είναι κάτι ουσιαστικό για να υποστηρίξουμε τι επιχειρήσει μας και να τι προστατεύσουμε από τι καταχρήσει και έπρεπε να, υπάρχει να δώσει μεγαλύτερη βεβαιότητα στι επιχειρήσει μα Το ίδιο ισχύει και για τι δημόσιε συμβάσει, το ίδιο ισχύει και για τι διαπραγματεύσει για την TTIP. Εσεί, ε, κύριε ε, Υπουργέ αναφερθήκατε στη δημοσίευση της Διαπραγματεύτικέ εντολή. Ναι, συνέβη αυτό. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το έγγραφο ήδη ήταν διαθέσιμο εδώ και ένα χρόνο. Έτσι λοιπόν δεν είναι και πολύ μεγάλη επιτυχία η δημοσιοποίηση αυτή. Επίσης θα μπορούσατε να εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία για να δώσετε όθηση με την Κομισιόν για την προστασία του Made in. Εγώ νομίζω ότι για το Made in χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Τελική Προεδρία ε, από πάρα πολλού παραγωγού και σε χρόνια ε, θεωρείται ότι ήταν η μεγάλη του ελπίδα και εγώ νομίζω ότι πραγματικά χάσατε αυτή την ευκαιρία. Εμείς ε, βασιζόμαστε σε εσάς και νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει και την ευθύνη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για τους... Ε, ε, ευχαριστώ πολύ για τις απόψεις σας σήμερα το πρωί που μας ε, εκθέσατε. Ένα θέμα θα ήθελα να μου για τα επίμαχα ορικτά. Βλέποντας το υπό το, την TTIP βρίσκεται κατά το ίμιση και μετά υπό την πρότασή σας η TTIP ζητεί να σταματήσει ή να αποσυρθεί το θέμα των επίμαχων ορυκτών. Η άλλη πλευρά ζητεί μεγαλύτερη δράση. Είναι λοιπόν επίμαχο ζήτημα. Ουσιαστικά θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπορική πολιτική μας για να δώσουμε συνέχεια στην πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θέλουμε να προασπίσουμε παγκόσμια. Και νομίζω ότι η τεράστια πλειοψηφία ε, ζητεί δεσμευτική κάμετρα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι εθελοντικού χαρακτήρα μέσα. Θα έχουμε και μια κρόση στο Ευρωκοινοβούλιο λίγο αργότερα σήμερα το πρωί για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να μου πείτε ποιε είναι οι απόψει στο Συμβούλιο. Βλέπετε κάποιο περιθώριο για δεσμευτικά μέσα και εργαλεία και όργανα και όσον αφορά την αλυσίδα ε, τροφοδότησης με αυτά τα ορυκτά θα ήθελα την άποψή σας γι' αυτό. Σε ευχαριστώ. Και εγώ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα όσον αφορά τις ε, ιδιωτικές δυνατότητες ε, επιδιαιτησίας ε, ε, θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Ταυτόχρονα όμως κάποια, κάποιοι υπέρμαχοι αυτού του μέσου στον Καναδά ή ε, στο, ΣΥΣΥΠΑ ε, ανελέητα υπονομεύουν αυτή τη δυνατότητα. Τι θα γίνει αν υπάρξει μικρότερο πλαίσιο, θα υπάρχουν λιγότερες επενδύσεις. Μέχρι σήμερα ήταν φραγμός ε, για τις επενδύσεις αμφωτέρωθεν του Ατλαντικού Ήδη σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη διασύνδεση και με τον Καναδά και με τη ΣΥΠΑ στο πεδίο επενδύσεων. Εκεί που έχετε δίκιο είναι ότι δεν μπορεί κανείς να πει ότι οι εθνικές και διμερείς ε, ε, συμφωνίες ESDS ε, είναι οι πιο λογικές. Δεν θα ήταν όμως λογικό να πει κανείς αυτές οι ρυθμίσεις, αυτές οι συμφωνίες είναι συμφωνίες του 20ου αιώνα όταν δεν ήταν τόσο αλληλένδετη η παγκόσμια οικονομία και αν τώρα το, προχω... το θέλουμε να το προαγάγουμε αυτό θετικά στο μέλλον, θα πρέπει να υπάρχει σαφέστατη δυνατότητα εμπλοκής ε, ε, παγκοσμία... παγκόσμιας επιδιαιτησίας ή ε, δικαστηρίων που θα έχουν διεθνώς την αρμοδιότητα αυτή. Ευχαριστώ. Πρόκειται για το χρονικό μιας αυτοκτονίας. Ε, δεν φταίτε εσείς, ε, οι κανόνες είναι που δεν λειτουργούν. Εσείς ε, μας παρουσιάσατε το θάνατο ενός οικονομικού συστήματος. Οι άλλοι είναι πιο έξυπνοι από εμά, τα καταφέρνουν καλύτερα και εγκαρασπίζονται τον εαυτό τους. Εμείς δεν τα καταφέρνουμε για την και για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, για τα πάντα για τα μέσα εμπορική άμυνα, εσεί ε, μα παρουσιάσετε με εικόνα ότι άλλοι προστατεύουν τα συμφέροντά του ε, ταχύτατα, προστατεύουν τα συμφέροντα των παραγωγών του και εμεί αντίθετα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρόλο τη δική σα και δική μα καλή θέληση, γιατί οι περισσότερε ε, χώρε υπερασπίζουν αυτόν που παράγει αλλού, εισάγουν στην Ευρώπη και πολλούν ξένα προϊόντα. Έτσι λοιπόν εδώ τι κάνουμε, παραδιδόμαστε. Ε, εσείς και εγώ πάμε έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ε, θα παρακολουθούμε στον υπόλοιπο κόσμο και θα πούμε είναι ανίκανη η Ευρώπη και είναι υπηρέτης αυτών που παράγουν αλλού. Εγώ δεν παραδίδω με το αντίθετο. Αυτό θα μας έλειπε, αλλά ε, το αποτέλεσμα είναι μηδέν, αλλά όχι από κακή βούληση, παρά τις ψήφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά γιατί αυτή η Ευρώπη είναι οικοδομημένη στα συμφέροντα άλλων. Σας ευχαριστώ γιατί μου επιβεβαιώσετε την ε, ιδέα αυτή, ότι τελικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ε, Κύριε όταν ρώτησα νωρίτερα για το ε, τι μπορεί να γίνει. Βεβαίως και ξέρω ποια είναι η θέση του ECR. Η έκθεση τώρα του εκπροσώπου της Προεδρίας είναι επικοδομητική, είναι σημαντική και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά στην κατεύθυνση αυτή. Τώρα για να μιλήσουμε για το ECR. Ξέρετε ότι το ECR ιδιαίτερα δίνει σημασία να εξεταστούν σε σχέση με το TTIP οι e κίνδυνοι Βεβαίω, κάθε τέτοιο βήμα μπορεί να σημάνει εντατικοποίηση του ανταγωνισμού. Υπάρχουν ευκαιρίες λοιπόν, όπως και υπάρχουν κίνδυνοι. Πρέπει λοιπόν πάνω απ' όλα να εκμεταλλευτούμε τι ευκαιρίες, αυτό σημαίνει πολιτική και αν δώσουμε προσοχή σε αυτό θα κερδίσουμε, θα είμαστε εμείς κερδισμένους. Εάν δούμε παραδείγματι τι διμερεί σχέσει τη Γερμανία με τι ΗΠΑ. Η Γερμανία έχει μεγάλο ε, πλεόνασμα στο εξαγωγικό της ισογυζύγιο προς τις πολιτείες Για δε τα διαιτητικά δικαστήρια. Βεβαίως πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει να κάνει και με την προστασία της ε, κρατικής κυριαρχίας και με την ασφάλεια των επενδύσεων. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι με την ασφάλεια δικαίου μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα και διασφάλιση των επενδύσεων. Και σε αυτό, σωστά είπατε κύριε ε, Πρόεδρε, ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στα σημεία αυτά που έχουν κέρια σημασία για τα διαιτητικά δικαστήρια. Γιατί καθοριστικός προς την TTIP δεν είναι η ανάπτυξη του ελεύθερου εμπορίου, αλλά η οπτική από την οποία θα δούμε τις επενδύσεις στην Ευρώπη, δηλαδή η Ευρώπη ως πόλος έλξους επενδύσεων. Εδώ θα πρέπει να είμαστε θέση να διαφυλάξουμε επενδύσεις με μεγάλα ποσά που θα έρθουν και εάν θέλουμε να περάσουμε αυτές τις ε, συμφέρουσες σχέσεις πρέπει να παραμείνει η πρόταση αυτή στην έκθεση και να προωθηθεί ακόμη περισσότερο και θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην ε, ε, παραπομπή σε ιδεολογικές διαφορές στην έκθεσή σας ή ιδεολογική τάφρος. Θέλετε να μας πείτε ακριβώς ποιες είναι οι τόσο μεγάλες διαφορές που χαρακτηρίζονται και ως τάφροι. Ποια είναι τα κράτη αυτά δηλαδή που διαφοροποιούνται πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ροδρίγες. Ε, σε ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να προσθέσω τη φωνή μου στα συγχαρητήρια προς την Ιταλική Προεδρία και να ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία της ενώπιών μας. Θα ήθελα να υποβάλω τρεις σκέψεις. Πρώτον, Μπορείτε να συγκεκριμενοποιήσετε περισσότερο πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί ο εξυγχρονισμός των μέσων εμπορικής άμυνας και ποιο χρονοδιάγραμμα θεωρείτε πιο σκόπιμο. Όλοι οι βιομηχανικοί και επιχειρησιακοί τομείς μας λένε ότι έχουν δυσκολία να ανταγωνιστούν σε τρίτες χώρες όπου χρησιμοποιούνται αθέμητες πρακτικές, κατά δηλαδή του ελεύθερου εμπορίου. Δύο, δεύτερο, εξακολουθώ να βλέπω ότι λείπουν προοπτικές ε, για το μέλλον για ένα πιο έντονο ρόλο της Λατινικής Αμερικής στην εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η εκτίμησή σας. Και τέλος, με ανησυχεί πολύ η στρατηγική παγκοσμίου εμπορίου της Κίνας και σε σχέση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον βραδύ ρυθμό και για τη δυνατότητα να υπογραφούν συμφωνίες ε, ευρύτερης εμβέλειας που να προστατεύουν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πείτε μου ποια είναι η άποψή σας. Ποια θα πρέπει να είναι η απάντηση της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν την κατάσταση. Ε. Πολύ γρήγορα για ε, και για το να απαντήσω και στον κύριο Σελβίνη και στους μίλησαν για το λογικό ρήγμα. Εγώ τι προσπάθησα να κάνω σε αυτή την Προεδρία, να αποφύγω, να χρησιμοποιήσω αυτό το γραφειοκρατικό επίσημο τόνο που χρησιμοποιείται συνήθως και είναι το εξή. Δεν καταλήξαμε σε συμβασμό, αλλά όλοι θέλουμε να συνεχίσουμε να συζητάμε για την επίτευξη κτλ. Απαντώ λοιπόν και σε εσά. Ο συμβιβασμό υποαυτήκε δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί γιατί το ίμιση των χωρών θεωρούν με σαφήνεια ότι η υιοθέτηση μέσων μπορούμε να, με τα οποία μπορούμε να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας ε, είναι προτεξιονισμός, προστατευτισμός. Εδώ και εγώ συμφωνώ με τον κύριο Σελβίνη. είναι η αυτοκτονία της ε, ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής. Αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι το να έχουμε μέσα εμπορικής άμυνας είναι ο τρόπος για να μπορούμε να έχουμε και μεγαλύτερο άνοιγμα, αλλά ε, συνεχίζουμε να μένουμε σε διάφορες ιδεολογίες ε, λέγοντας ότι είναι αφηρημένο φαινόμενο παγκοσμιοποίηση και όχι συγκεκριμένο φαινόμενο όπου εδώ μετρώνται τα συμφέροντα ε, των χωρών σε επίθεση σε άμυνα, όπω κάνουν οι ανταγωνιστές, Εμεί ε, πηγαίνουμε κατευθείαν να χτυπήσουμε το κεφάλι μα στον τοίχο. Συμφωνώ απόλυτα λοιπόν, ο στόχο της Προεδρίας μας δεν ήταν να φτάσουμε σε μεσμό, δεν ήταν δυνατό. Εγώ δεν μπορούσα να φεύγω τα πάντα από το μηδέν, αλλά τουλάχιστον αυτό, να σα πω ξεκαθαρά πώς έχουν τα πράγματα. Στο πλαίσιο του εγγράφου στρατηγικής κομισιόν ε, που ζητήσαμε, α δούμε εκεί τι ακριβώ θέλουμε να κάνουμε για το εμπόριο. Εγώ που διαφωνώ τώρα κάθετα με τον κύριο Σελβίνη ότι η στρατηγική δεν μπορεί να είναι μόνο στρατηγική άμυνα, γιατί η ανάπτυξή μας εξαρτάται από την πρόσβαση στην αγορά. Έτσι λοιπόν, ε, ωραία μου λέτε πρέπει να είμαστε πιο ισχυροί στην άμυνα αλλά αν δεν υπάρχει και μια πολιτική όπου εμείς δεν έχουμε πρόσβαση στην αγορά τότε με τον ίδιο τρόπο θα έχουμε ε, μια αργή πτώση. Έτσι λοιπόν, ας μην ε, κάνουμε εδώ ε, κάποιες χειρονομίες πολύ έντονες, αλλά ας ε, κάνουμε τις κατάλληλες ενέργειες για να έχουμε αμήνα αλλά και επίθεση. Γιατί δεν μπορούν να σκεφτούν κάποιοι ότι το μόνο που θα κάνουμε είναι να βάλουμε εμπόδια, θα πρέπει να σπάσουμε και κάποιο τοίχο. Τώρα για το Made in. Δεν είναι αρμοδιότητα της, του Συμβουλίου Εμπορίου. Το Made in είναι θεμελιώδες. Εγώ είχα κάνει τότε τη μάχη, είχα δώσει τη μάχη με την Confindustria και είχαμε φτάσει απόσταση μία ψήφου. Δεν ολοκλήρωσε, δεν ολοκληρώθηκε βέβαια το εξάμεινο. Εγώ συνεχίζω αυτή τη μάχη μέχρι τέλους. για τη Λατινική Αμερική, την Κίνα και τι επενδύσει. Η Λατινική Αμερική είναι η εξή κατάσταση. Όλο ένα κλείνεται περισσότερο το Μερκοσούρ. Αφήσουμε την Ελληνική. Η Βραζιλία αυξάνει ε, τους δασμούς. Τώρα πρέπει να δούμε τι κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, δηλαδή, συμμαχία με τις χώρες που δέχονται τους κανόνε, Χιλή, Περού, Κολομβία, Μεξικό, Κεντρική Αμερική αν εμείς ε, κάνουμε κάτι τέτοιο θα οφήσουμε και τη Βραζιλία ε, στον ανοιχτή, αν έχουμε την κριτική μάζα. Αυτή πρέπει να είναι στρατηγική επίθεση που πρέπει να ακολουθήσουμε, γιατί πρέπει να υπάρχει και ικανότητα βέβαια από τη Δύση να την ε, θέσει σε εφαρμογή αυτή τη στρατηγική Κίνα. Πρέπει να προχωρήσουμε με τις επενδύσεις έχουμε ένα μέσο που θα μπορούσε να είναι καινούριο. ρόλος της Κίνας στον Παλί ήταν κάτι καινούριο στα συμπεράσματα του ΠΟΕ. Έχει απομακρυνθεί από τις άλλες χώρες BRICS και υποστήριξε, είχε μια θετική υποστήριξη. Η διάσκεψη του Πεκίνου, όπου εκεί η Ινδία και η Κίνα συμφώνησαν για το κλίμα και για τεχνολογικά αγαθά, υπάρχει ένα μήνυμα που μας δίνει ότι κάπως η Κίνα αρχίζει να αλλάζει αυτή τη στάση Δηλαδή περισσότερο επικοδομητική φαίνεται η Κίνα. Πρέπει να το έχουμε αυτό κοντανού και να μετρήσουμε τις επίσημες πρόοδους. Γιατί ακόμα και εμεί δεν κατορθώσουμε ε, να είμαστε ενωμένοι, όπω παραδείγματο χάρη στην περίπτωση των Βοτελτικών, είδαμε ότι δεν είναι έτοιμη η Ευρώπη να αντιπαραταχθεί. Πρέπει να βρούμε εναλλακτική στρατηγική. Τώρα για τα ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες, ε, αύριο στην ημερησία διάταξη της ε, TPC ε, υπάρχει το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των κρατών μελών. Ε, τώρα, για το αν θα έχουμε υποχρεωτικό ή ακούσιο χαρακτήρα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εγώ συμφωνώ ε, η εμπορική πολιτική να ευνοήσει διάδοση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά θα πρέπει και να μην οικοδομήσουμε μηχανισμού που κατόπιν είναι πολύ δύσκολο να του διαχειριστούμε και θα ζημιώνουν τη βιομηχανία χωρί να προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό περισσότερο είμαστε υπέρ του εκούσιου χαρακτήρα παρά του υποχρεωτικού. Σα ευχαριστώ. Yeah, thanks a lot, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ που ήρθατε για άλλη φορά. Και ευχαριστώ που αγωνίζεστε για την πολιτική μας του διεθνού συμπορίου και κάθε επιτυχία εύχομαι. Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι περνάμε στις ψηφοφορίες τώρα και καταρχήν 16 δασμολογική κάλυψη προϊόντων σημερινού Εκουαδόρ. Συζητήσαμε χθες για αυτό το θέμα και κατά τούτο είναι όλα πλέον σαφή και ξεκάθαρα και μπορούμε να ψηφίσουμε. Έχουμε καταρχήν την συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 της Ενωτικής Αριστεράς και των Πρασίνων, Γκουε και Πρασίνων. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για να είμαστε βέβαιοι για το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τον συμβιβασμό 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Σαφές το αποτέλεσμα. Και περνάμε στη συνέχεια στην τροπολογία 20. Υπέρ, κατά, αφοχές, απορρίφθηκε. Τροπολογία 21. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Πάμε στην τροπολογία 22, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τροπολογία 8, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Πάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 2 υπέρ συμβιβαστική κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 15, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα τώρα της 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Και πάμε τώρα. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε για το κείμενο αυτό, δηλαδή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας από το ΕΛΚ παραπάνω ψηφίζει. Πρέπει ένας να αφαιρέσει την ψήφο του. Εντάξει, ωραία, πέρας ψηφοφορίας τώρα. <coughs> με 34 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε η πρόταση. Και θα περάσουμε τώρα και θα ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Και εδώ πάλι ηλεκτρονικά και άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα 35 ψήφοι υπέρ. Εγκρίθηκε λοιπόν το κείμενο του ψηφίσματος. Παρέμβαση εκτός μικροφώνου. Να έχουμε και μια πρόσθετη αποχή. Εντάξει, δεν πειράζει. Η πρόταση λοιπόν της Επιτροπής εγκρίθηκε υπ' αυτή τη μορφή και σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι ο, η και τα προϊόντα του δεν θα βρεθεί σε ένα κενό. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 17. Ο Χέλμουτ, Χέλμουτ Σόλτς παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προτείνω να ξεκινήσουμε αμέσως με τις διαπραγματεύσεις ε, για αυτό το θέμα ή μήπως πρέπει να ψηφιστεί πρώτα. Αν θέλετε μπορεί να γίνει. Ε, Πρόεδρε, Νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεκινήσει κάποια άμεση διαπραγμάτευση, ούτως ή άλλως. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να ξεκινήσει κάποια διαπραγμάτευση. Διότι έγινε δεκτή η πρόταση τη Επιτροπή, Μετά θα πάμε στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο, το δυνατόν πιο νωρί. Και αν κερδίσουμε πάλι δεν θα υπάρξει τριμερή διάλογο αν εγκριθούν οι προτάσει του κυρίου Σόλτ, τότε θα υπάρξει τριμερή διάλογο, όχι τώρα. Και αυτή τη νομική άποψη έχω και εγώ Χέρμουντ Σόλτ, γιατί δεν εγκρίθηκε κάποια τροπολογία σου και έτσι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει αναλύωτη. Και δεν θα, υπήξε, δεν θα υπάρχει ε, ανάγκη να διαπραγματευτούμε. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα ποια είναι η συγκεκριμένη θέση του Συμβουλίου επ' αυτού. Δηλαδή, αν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα, τότε θα έχουμε πάλι την ίδια κατάσταση τον Ιανουάριο. Γι' αυτό θα έλεγα τουλάχιστον να βρούμε, να διαπιστώσουμε ποια είναι η θέση του Συμβουλίου επ' αυτού. Uh, Μάλιστα, είναι απόλυτα σαφέ. Αν από το Συμβούλιο υπάρξει κάποια τροπολογία σχετικά, τότε θα πρέπει το δυνατόν ταχύτερα να κάνουμε μια έκτακτη συνεδρίαση για να αποφασίσουμε εμεί. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια επισήμανση ή κάποια προαναγγελία ότι το Συμβούλιο θα άλλαζε κάτι. Το Συμβούλιο εκπροσωπείται εδώ σήμερα. Ναι ή όχι. Ναι, ήταν εδώ πριν. Μάλιστα, αλλά τι γίνεται τώρα. Μπορεί να πει ότι είναι υπέρ, ήταν υπέρ. Δεν αναμένω εγώ κάποια αλλαγή, κάποια τροπολογία να κατατεθεί. Αλλά να ξέρουμε, αν θα υπάρξει τροπολογία θα πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι θα υπάρξει κάποια τροπολογία από το Συμβούλιο. Λοιπόν, πολύ καλά. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο σημείο 17. Χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων για τη δημοκρατία της Μολδαβίας. Ψηφίζουμε. Περνάμε στην τροπολογία 7 της κυρίας Λεπέν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Μάλιστα. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 3 υπέρ σεγίγεν κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε και περνάμε τώρα να ψηφίσουμε την τροποποιημένη ή μη τροποποιημένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ αυτής παρακαλώ ναι ναι σαφές συγγνώμη ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε βέβαια σωστό ζητώ συγγνώμη άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 34 υπέρ και 5, 5 ψήφοι εναντίον, 2 αποχές. Και για το νομοθετικό ψήφισμα τώρα πάλι ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και εδώ πάλι 34 ψήφοι υπέρ, 4 εναντίον και 3 αποχές. Εγκρίθηκε και αυτή η πρόταση. Μάλιστα, συγχαρητήρια προς τον εισηγητή. Και περνάμε τώρα στη συνέχεια στο σημείο 18 της ημερήσιας διάταξης. Εδώ πρόκειται για την πρόταση ψηφίσματος για το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων συν διευρυμένο έχουμε τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε μια κατεξουσιοδότηση πράξη που θα ασκήσουμε επικρίσεις ή θα εκφράσουμε την ένσταση και αντίρρησή μας. Και έχουμε δύο τροπολογίες επ' αυτού στο ψήφισμα που πρέπει να ψηφιστούν πρώτα. Η τροπολογία 1 λοιπόν πρώτα, υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε και τώρα θα ψηφίσουμε το ψήφισμα στο σύνολό του ηλεκτρονικά βέβαια και άρχεται η ψηφοφορία επ' αυτού Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα άλλη μια ψήφος υπέρ, εντάξει 12 λοιπόν υπέρ αλλά 26 εναντίον και τρεις αποχές. Απορρίφθηκε λοιπόν το ψήφισμα. Απορρίφθηκε. Με άλλα λόγια, τι σημαίνει αυτό. Η κοινοβουλευτική μας επιτροπή δεν θα έχει ψήφισμα που θα κατατεθεί στην Ολομέλεια. Υπάρχει φυσικά η δυνατότητα με 40 υπογραφές 40 ε, ε, ευρωβουλευτές ή μια κοινοβουλευτική ομάδα να ζητήσουν να κατατεθεί αυτό το αίτημα στην Ολομέλεια. Και περνάμε στο επόμενο σημείο, στο 19 που πρέπει να ψηφίσουμε. Είναι η ρύθμιση για πρόσβαση στην αγορά <clears throat> για την Κένια προϊόντων της Κένιας. Έχουμε μία ψήφιση που θα γίνει και θα γίνει ηλεκτρονικά η ψηφοφορία αυτή. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία αυτή. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 37 υπέρ. Μάλιστα, 37 υπέρ. 2 εναντίον και μία αποχή. Και έτσι ολοκληρώσαμε τον γύρο ψηφοφοριών για σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστώ θερμά. Δύο λεπτά θα κάνουμε διάλειμμα για να προετοιμαστούμε για την ακρόαση που ακολουθεί. Α, So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmen Sie denn langsam... Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε με την ησυχία Ja, liebe Kolleginnen und Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, περνάμε τώρα στο σημείο 20 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για την ακρόαση, για το εμπόριο ορυκτών προερχομένων από περιοχές συγκρούσεως και υψηλού κινδύνου. Καλώς ήρθατε στην σημαντική αυτή ακρόαση. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί εδώ και καιρό στην, στο νομοθετικό μας έργο. Ξέρετε ότι προσπογράφουμε τις ευρωπαϊκές αξίες και ταυτόχρονα θέλουμε οι πρώτες ύλε που αξιοποιούμε σε πολλούς τομείς να αξιοποιούνται, να προκύπτουν έτσι, να εξορίσονται έτσι, ώστε να μην παραβιάζονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι γνωστή αντιπαράθεση σε σχέση με τη σχετική νομοθεσία στα Ηνωμένα Έθνη, στις Ηνωμένε Πολιτείες, η οποία επιδιώκει αντίστοιχους στόχους, ιδιαίτερα στην περιοχή των Μεγαλών Λιμνών και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που, που θα έπρεπε να έχει προχωρήσει εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία θα αναλύσουμε παράλληλα με αυτή την ακρόαση και θα μπορέσουμε έτσι να έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις διάφορες πτυχές και όψεις του προβλήματος. Πριν δώσω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Βίνκλερ, εισηγητή μας, Θέλω να καλωσορίσω τους πυρογνώμονε και προσκεκλημένους μας, ειδικού στους διαφορούς τομείς. Θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερω για την παρουσία τους εδώ και την ευκαιρία να μας ε, διαφωτίσουν με τις γνώσεις τους. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 12.30. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε ο καθένας να είμαστε σύντομοι και συνεκτικοί. Παρακαλώ λοιπόν ως εκ τούτου και τους ειδικού μας να περιορίσουν τις ομιλίες τους στις, στα 8 λεπτά, 8 λεπτά χρόνο ομιλίας. Έχουμε δύο γύρους παρουσιάσεων και την ευκαιρία βέβαια για συζήτηση, την οποία ιδιαίτερα θα ήθελα να αξιοποιήσω και θα, θα είναι όσο το δυνατόν πιο παρατεταμένη ανάλογα με την διάρκεια των ομιλιών και παρουσιάσεων. Αλλά πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Βίνκλερ, εισηγητή μας. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φιλοξενούμενοι. Θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω δύο λόγια, να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και τους υπαλλήλους που διοργάνωσαν αυτή την ακρόαση σήμερα, που είμαι πεισμένος ότι θα είναι πάρα πολύ γόνιμη και θα μας δώσει πολλές πληροφορίες. Σας ευχαριστώ επίσης σε εσάς πολιτικές ομάδες και σκιώδεις εισηγητές, κοινοβουλευτικές ομάδες και σκιώδεις εισηγητές για αυτή τη διαδικασία μέσα στην οποία διαπραγματευτήκαμε, συζητήσαμε και καταλήξαμε σε μια κοινή επιτέλους θέση για τη σύνθεση των πάνελ και των πραγματογνωμόνων που θα παραστούν σήμερα ανάμεσά μας και πιστεύω ότι στρεφόμενος στο θέμα τώρα το ίδιο επί της ουσίας είναι προφανές λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η Ευρωβουλή, το Ευρωκοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει ένα ψήφισμα και την τοποθέτησή του για το θέμα των ε, επίμαχων αυτών ορυκτών και το γεγονός ότι ανταποκρίθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπέβαλε την πρότασή της για κανονισμό σε σχέση με αυτό το θέμα, είναι πλέον σαφές ότι πρέπει να εξετάσουμε με πολύ υπεύθυνο τρόπο, με μεγάλη ευθύνη τα ζητήματα. Ο στόχος είναι σαφής και με συνένεση επετέχθη. Πρέπει να καταφέρουμε να διαρρήξουμε τον δεσμό σε σχέση με την προέλευση από επίμαχες περιοχές και την επεξεργασία και εκμετάλλευση αυτών των ε, ορυκτών. Πώς θα γίνει αυτή η δράση θα το δούμε. Νομίζω το καλύτερο από πλευράς μου θα ήταν τώρα να αφήσω περισσότερο χρόνο στους ε, πραγματογνώμονες και να ολοκληρώσω εδώ. Ολοκληρώνω εδώ και αδειμονώ και προσβλέπω στο τι θα μας πούν οι επαΐοντες. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βίνκλερ. Και ξεκινάμε τον πρώτο γύρο τώρα με τις πανεβάσεις των πραγματογνωμόνων που θα αντιμετωπίζουν το θέμα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα διεθνές αριθμιστικό πλαίσιο. Πρώτα απ' όλα έχω την τιμή να δώσω τον λόγο στον κύριο Τάιλερ Γκίλαρντ, νομικό σύμβουλο στην, ε, στον ΩΣΑ, στην, ε, ε, στο τμήμα επενδύσεων και η αρμοδιότητά του είναι αυτή. Έχετε τον λόγο κύριε Γκίλαρντ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Με χαρά έρχομαι να σας μιλήσω σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη τιμή που έχω την ευκαιρία να απευθύνομαι στην Επιτροπή σας για το σημαντικό αυτό θέμα των ε, περιοχών που πλήττονται από ε, συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου. Ονομάζομαι λοιπόν Tyler Gillard, είμαι νομικός σύμβουλος στον ΩΣΑ για τα θέματα αυτά και θα ήθελα να αφαιρθώ σήμερα στο κύριο μέσο που έχουμε στη θέση μας, δηλαδή τις κατευθυντήρες γραμμές του ΩΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού με ορυκτά από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου για να σας αναφέρω το πώς σχετίζονται αυτά όλα με το θέμα μας. Από το 2009 έχει ξεκινήσει ο ΣΑ προσπαθώντας να αναπτύξει υπεύθυνα ε, μέσα ε, εξόριξης ορυκτών ε, κατά τρόπον ώστε να μην επιτείνονται τα προβλήματα και να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στο αντικείμενό μας που είναι χώρες ΩΣΑ και μη ΩΣΑ, την κοινωνία των πολιτών, το και κοινωνίες εμπειρογνώμονες. Όλα αυτά τα λέω διότι έχουμε ιδιαίτερα δώσει έμφαση στη συνεργασία με τις αφρικανικές χώρες. Οι κατευθυντήρες γραμμές περιγράφουν τι είδους ε, μέσα θα πρέπει, μέτρα θα πρέπει να εισαγάγουν οι χώρες ώστε να εξασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να αποφεύγεται δηλαδή η αξιοποίηση συγκρούσεων. Έχουμε έχουν υιοθετεί από 43 χώρες, τις χώρες του ΟΣΑ είναι νέα ακόμη δηλαδή, αυτές οι συστάσεις. Πρόκειται για σύσταση του ε, Συμβουλίου του ΟΣΑ με προσπάθεια για προώθηση αυτών των κατευθυντηριών γραμμών γενικότερα και εφαρμογή τους. Όλα τα κράτη-μέλη που προσυπέγραψαν λοιπόν αυτές ε, τις συστάσεις και το σχέδιο κανονισμού αποτελεί μια ευκαιρία για πρωτοπορία στο σημαντικό αυτό θέμα. Με χαρά βλέπουμε ότι το σχέδιο κανονισμού στηρίζεται στις αρχές της δέουσας επιμέλειας και τις κατευθυντηρίες μας γραμμές. Τι σημαίνει εδώ δέους επιμέλεια. Σημαίνει ευφυή, συνεχή διαδικασία. Οι επιχειρήσεις, τα κράτη ορίζουν συστήματα διαχείρισης, εντοπίζουν τους κινδύνους ε, που μπορεί να προκύπτουν από περιοχές σύγκρουσης, ορίζουν προδιαγραφές ε, για την αλυσίδα προμήθειας, ε, και ελέγχουν την τήρησή τους. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με τέσσερα βασικά βήματα. Θα ήθελα να σας εξηγήσω τι ακριβώς είναι το πεδίο αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής από το ορυχείο έως τον καταναλωτή. Είτε πρόκειται για χιτήρια, είτε πρόκειται για καταστάσεις τήξης, είτε πρόκειται για τα ορυχεία, για τη διαχείριση, υπάρχει υποχρέωση για την παρακολούθηση και τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πώς όμως θα τηρηθούν αυτές οι ευθύνες θα εξαρτηθεί από τον, ε, από τον τρόπο στον οποίο, από τη θέση που έχει ο καθένας αυτήν την αλυσίδα προμήθειας. Και εμείς προσφέρουμε πρόσθετες κατευθυντηρίες γραμμές για τη δέουσα επιμέλεια από το ανώτερο σημείο, δηλαδή το ορυχείο, της αλυσίδας παραγωγής μέχρι και το χειριτήριο ή την εγκατάσταση τήξης ε, και μέχρι και το κατώτατο σημείο, τον καταναλωτή δηλαδή, το κατώτερο της αλυσίδας κατευθυντήριες γραμμές ειδικέ δηλαδή. Γιατί ο κάθε ένας από τους ε, παράγοντες αυτούς μπορεί να έχουν διαφορετική θέση, επιρροή, επίδραση ή απόδοση στην υπόθεση αυτή. Άρα μπορεί ε, να είναι δυνατόν να καταστεί γνωστό το ορυχείο προελεύσεως, η αλυσίδα της μεταφοράς του προϊόντος, η ποιοτική αξιολόγηση της θέσεως του ορυχείου, στο ανώτερο επίπεδο, της, στο αρχικό επίπεδο της αλυσίδας, ενώ στο κατώτερο επίπεδο, στο τελικό δηλαδή, πρέπει να γνωρίζει κανείς από ποιο χιτήριο πέρασε, από ποια εγκατάσταση τήξης. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει απολύτω μέχρι και το ορυχείο προελεύσεω του προϊόντος ο τελικός καταναλωτής, αλλά το χιτήριο πρέπει να το γνωρίζει. Ε, έλεγχη λοιπόν που σημαίνουν έλεγχο για το χιτήριο και την εγκατάσταση τήξης, ε, που είναι κέριο σημείο, μόνο λοιπόν για αυτούς. Με 500 χιτήρια και εγκαταστάσεις τήξης καλύπτουμε το 95% της παραγωγής, των τριών τι όπως τα ονομάζουμε, δηλαδή κασίτερο, ε, βολφράμιο, ε, ταντάλιο και χρυσό, τα τρία τάφσιν χρυσός. Παρακαλουθούμε ως εκ τούτου την επεξεργασία των προϊόντων αυτών. Τα μέταλα και ορυκτά παρακολουθούνται ως τμήμα της αλυσίδας και γίνονται οι έλεγχοι. Πρόσθετες ε, προϋποθέσεις πέραν των χιτηρίων και καταστάσεων τήξεως ε, που προβλέπονται στις, ε, στα αιτήματα θα δυσκόλευαν ενδεχομένω με επικαλύψεις το έργο μας και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Για να έχουμε όμως καλύτερη εφαρμογή των κατευθυντηριών γραμμών Πιστεύουμε ότι θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει ότι όλες οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα προμήθειας που έχει να κάνει με ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων θα είναι τουλάχιστον υποχρεωμένες να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές της ε, δέουσας επιμέλειας στην ε, ε, καταγραφή, στις δηλώσεις τους για τα προϊόντα τους. Υπάρχει ένας μηχανισμός με ένα σχέδιο κανονισμού που μπορεί και το σχέδιο κανονισμού λέω θα μπορούσε να επεξεργαστεί περαιτέρω τις λεπτομέρειές του. Οι κατευθύνες γραμμές αφορούν όλα τα ορυκτά από κάθε περιοχή υψηλού κινδύνου ή συγκρούσεων ανά τον κόσμο. Οι κατευθυντήριε γραμμέ απαιτούν από τι επιχειρήσει να ακολουθήσουν τι αρχέ τη δέουση επιμέλεια, γιατί εδώ ακριβώ βρίσκονται οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι, δηλαδή τη χρηματοδότηση ένοπλων βίων συγκρούσεων, παραβιάσει ανθρωπινών δικαιωμάτων. Οι κατευθυντήριε γραμμέ όμω περιλαμβάνουν μόνο τις ε, ειδικέ προδιαγραφέ δέους επιμέλεια για τα τρία τι και το χρυσό που σα ανέφερα νωρίτερα, βολφράμιο, κασίτερο, ταντάλιο και χρυσό. Εδώ είναι το τελευταίο κομμάτι τη έκθεσή μα όπου γίνεται η αξιολόγηση του κινδύνου και μετά έχουμε τι ειδικέ προδιαγραφέ για τα τρία τάφ και το χρυσό με τι συμπληρωματικέ προδιαγραφέ δέους επιμέλεια που σα περιέγραψα. Το σχέδιο κανονισμού λοιπόν περιλαμβάνει μόνο πιστοποίηση για τα τρία τάφ και το χρυσό κασίτρο βολφράμιο, ταντάλιο και χρυσό, όπως έχει εστίσει το πρόγραμμά μας και δίνει λεπτομερείς προδιαγραφές για την αλυσίδα προμηθειών. Αλλά διαφέρει προς το εξής, ότι οι κατευθύνες γραμμές προτείνουν να τηρείται η σε επιμέλεια από τις επιχειρήσεις με τα πέντε βήματα που περιλαμβάνονται στις δικές μας ε, κατευθυντήρες γραμμές. Εάν χρειαστεί λοιπόν επιπλέον έλεγχος ή πιστοποίηση, από, τον, ε, από το σχέδιο κανονισμού για άλλα ορεικτά θα πρέπει αυτό να γίνει με βάση τις ανάγκες και τις τεχνικές προδιαγραφές που ε, θα επέτρεπαν ένα τέτοιο έλεγχο και εμείς είμαστε διαθέσει για να βοηθήσουμε. Πάντως ε, θα πρέπει οι, οι χώρες και οι επιχειρήσεις να ενημερώνουν. Ιδιαίτερα θέλουμε να βοηθήσουμε στην τήρηση σαφών διαδικασιών λογοδοσίας από επιχειρήσεις ε, του ΑΟΣΑ και της Αφρικανικής Υπήρου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προαγάγουμε την εφημερία της θέσης εργασίας, την τοπική ανάπτυξη και έχουμε μια επικοδομητική προσέγγιση στις κατευθυντήριες γραμμές, δηλαδή πρέπει ο κλάδος αυτός της εξόριξης σταδιακά να προσαρμοστεί στις κατευθυντήριες γραμμές, ε, και αναλόγως να προσαρμόσει τις αποφάσεις. Άρα, άμα κοιτάξει κατευθυντήριες γραμμές, είναι πολύ συγκεκριμένη η ε, ορολογία που χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί η υπεύθυνη συμπεριφορά των παραγωγών στην αλυσίδα παραγωγής. Δεν περιμένουμε 100% τέλεια ε, προσαρμογή και τήρηση της δέουσας προσοχής, γιατί δεν αποτελεί αυτή την εγγύηση της καλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των προδιαγραφών μας, αλλά θέλει μια καλή τυπή στη διαδικασία, η οποία θα φέρει αποτελέσματα στον χρόνο. Ευελιξία λοιπόν, που είναι απαραίτητη και ενσωματώνεται, ιδιαίτερα χρήσιμη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να μπορούν να επιδεικνύουν και αυτές τη δέουσα προσοχή, όπως οφείλουν να την επιδεικνύουν, αλλά προβλέπουμε και τη σχετική ευελιξία προς όφελός τους. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιοποιήσουν και τις πρωτοβουλίες που αφορούν περισσότερους εμπλεκόμενους και επιχειρήσεις για να επιτελούν καλύτερα το έργο τους επί, υπό την έννοια της δέουσας επιμέλειας. Οι κατευθυντηρίες γραμμές, ναι, ξέρω ότι τελειώνει ο χρόνος μου, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πάντως τη χάνουν υποστήριξη και από τη Γενική Συνέλευση των Εθνών και από το Συμβούλιο Ασφαλείας, από χώρες όπως και η ακτή του Ελεφαντοστού, και χρηματοδοτείται πρέπει να πω από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι σημαντικός χορηγός ε, του προγράμματός μας με την κατάρτιση που προσφέρουμε, με τη βελτίωση των δεξιοτήτων, με την ε, επιτόπου ε, εμπλοκή μας και ελπίζω ότι θα είναι επιτυχές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Επόμενο εμπειρογνώμονα είναι ο κύριο Μπόντζα Μαλάση από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, πρόεδρος της ε, Κοινωνίας των Πολιτών ε, του Νότιου Κιβού. Παρακαλώ. Αξιότιμε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι παρεμβαίνω εκ μέρους ε, του πληθυσμού του Τιμπούντα που, και ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο που μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη θέση μας για την πρόληψη ε, και την καταπολέμηση των ενόπλων σειράξεων στη χώρα μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί την διαδικασία ε, της αναδιάρθρωσης του Κογκό για τον εκδημοκρατισμό, την καταπολέμηση της ατιμορρησίας, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι όσο ε, τόσο τα, όσο δεν λύνονται τα σημαντικά θέματα σε σχέση με τις τη σειράξεις, οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Και μεταξύ των τιών υπάρχει και η παράνομη εκμετάλλευση των πρώτων υλών που τροφοδοτούν τη σύραξη. Το πλαίσιο είναι το εξή επιτόπου. Καταρχήν έχουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκαλούνται από αυτή την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και αυτό φυσικά γίνεται και με την εμπλοκή στρατιωτικών σε τρία επίπεδα. Καταρχήν έχουμε τους, του στρατιώτες του τακτικού στρατού, έχουμε τις ένοπλες ομάδες που ασκούν τον έλεγχο ε, στις στα ορυχεία. Ε, επίσης, ε, παράνομη φορολόγηση γύρω από την τοποθεσία αυτών των ορυχείων στην ανατολική περιοχή του Κογκό και επίσης ε, στην επικράτεια της Αμπούντα υπάρχει ένας νέος τρόπος εκμετάλλευσης του χρυσού ε, με κάποια μηχανήματα. Για κάθε τέτοιο μηχάνημα ο διοκτήτης καταβάλει 2.000 δολάρια στο στρατιωτικό και ε, κατόπιν ε, πληρώνεται, καταβάλλεται φόρος 800 δολάρια και υπάρχει και συνενοχή του τακτικού στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας με τις ε, πολιτοφυλακές, με τις ένοπλες ομάδες και βρίσκουν, κάνουν κάποιες συμφωνίες με τις επιχειρήσεις προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση στις τοποθεσίες όπου ελέγχουν έχουμε μια τελευταία περίπτωση ε, μιας επιχειρήσης Kun Mining Group ε, με γαλλική και κινέζικη ηγεσία και κατόρθωσαν ε, το 2014 να λάβουν έγκριση από το στρατό και από τις τοπικές αρχές για να μπορούν να υπογράψουν μια συμφωνία με μια ε, πόλη, το φυλακή του Ριάν Μπόκι, ε, που ελέγχεται από τον Αλεξάνδερ Μωάμι. Έτσι λοιπόν ε, είναι δύσκολο οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να συνεισφέρουν ε, στην ειρήνη, στη λαϊκή δημοκρατία του Κογκό, γιατί υπάρχει πάντοτε αυτό το θέμα της εκμετάλλευσης των μεταλλευμάτων που πάντοτε θα τροφοδοτεί τις σειράξεις επιτόπου. Έχουμε, παραδείγματο χάρη, τα μεταλλεύματα ε, που παράγονται στη Σαμπούντα και στο Φίζι. Πρόκειται για μέρη που κυρίω ελέγχονται από αυτέ τι πολιτοφυλακέ ε, Ράιν Τομπόκι και πιστοποιούνται από τις αρχές, εξάγονται από τις αρχές ε, με το πιστοποίηση από ορισμένες τοποθεσίες της επικράτησης του ΟΚΟΥΜ και απλώς αυτό γίνεται για να μην σεβαστούν ε, την δέουσα επιμέλεια του ΣΑ που εμείς χαιρετίζουμε σε τοπικό επίπεδο. Είναι λοιπόν σημαντικό σαφή μέτρα να μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή για να βρούμε λύσεις. Έχουμε και τους πολίτες που πολλές φορές ε, αναγκάζονται να μετακινηθούν γιατί υπάρχει ε, σύγκρουση μεταξύ αυτών των ενόπλων ομάδων για να ελέγξουν τα ορχεία. Έτσι λοιπόν υπάρχει εκτοπισμός ε, του πληθυσμού. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα λάβει αυτά σοβαρά υπόψη και μέσω του Κοινοβουλίου σας έτσι ώστε ο πληθυσμός μας να μπορεί να ζήσει ειρηνικά. Στη Σαμπούντα υπάρχει μια νέα μορφή εκμετάλλευση του Χριστού στον ποταμό Ουλίντι και στον ποταμό Λουγκούλου με αυτές ε, τις μηχανές που σας ανέφερα. Αυτή ε, έχει οδηγήσει στην αύξηση των επιθέσεων. Κάθε τρεις μέρες έχουμε συγκρούσεις μεταξύ των αεροπλωμάτων για να ελέγχουν τις τοποθεσίες εξόρυξης. Και επίσης έχουμε και αύξηση του ιού του AIDS με αυτή την νέα μορφή ε, πριν αυτή την νέα μορφή ήταν στο 2% το AIDS, αλλά τώρα με αυτή την νέα εκμετάλλευση στις εμπούτες στο νοσοκομείο θα δείτε ότι το ποσοστό πέρασε στο 13% από το 2%. Έτσι λοιπόν μετά το τράκιο ε, θα έχουμε την εξαφάνιση του πληθυσμού. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα ε, υπάρχει και ο νόμος Ντοτ Φρανκ. υπάρχει μια εκστρατεία αμάβρωσης αυτού του νόμου γιατί έλεγαν ότι υπάρχει απώλεια θέσεων εργασίας ε, όμως εμείς πιστεύουμε ότι αυτός ο Αμερικανικός νόμος ε, έχει περισσότερα θετικά αποτελέσματα γιατί για πρώτη φορά ε, διαπιστώθηκε ότι εμπλέκονται και οι τοπικές αρχές και οι ενόπλες ομάδες στην εκμετάλλευση ε, των ε, μεταλλευμάτων και μάλιστα επειδή ο αρμόδιος θύμωσε πάγωσε την παραγωγή μεταλλευμάτων. Έτσι λοιπόν είδαμε θετικά αποτελέσματα δημιουργήσαμε κάποια, ε, κάποιες τοποθεσίες όπου μπορεί να πάει ο ντόπιο πληθυσμός, κάποια κέντρα όπου μπορεί να πάει και να καταγγείλει το τι βιώνει επί τόπου και δημιουργήθηκε μία μονάδα σε επίπεδο τακτικού στρατού ε, για να ελέγχει ε, αυτές τις τοποθεσίες. Και επίσης υπάρχουν και κάποια μέτρα να δημιουργούνται κοπερατίβες όμως, εμείς πιστεύουμε το εξής, μπορεί να πούνε επιχειρήσεις, ε, όχι υπάρχουν πάρα πολλές περιποθέσεις, όμως εμείς θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη έτσι ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε τέλος ε, σε αυτή την προβληματική της παράνομης εκμετάλλευσης ε, των μεταλλευμάτων που τροφοδοτούν τις σειράξεις. Δεν θα αλλάξει η κατάσταση εν μία νυχτή. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λάβει κάποια μέτρα που θα μπορούν να βελτιώσουν και την Αμερικανική νομοθεσία και καλούμε την να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ε, νομοθετική πρόταση για να καταπολεμήσουμε αυτή την παράνομη ε, τροφοδότηση των σειράξεων. Θέλουμε να έχουμε ε, συγκεκριμένες διώξεις κατά των μαφιόζικων των μαφιόζων και μιλάμε και για τη συμμετοχή ένοπλων ομάδων αλλά και του τακτικού στρατού Θέλουμε επίσης να υπάρξει από τις ε, επιχειρήσεις ε, ε, ότι θα τεθεί ο μηχανισμός εφαρμογή και δεν θα μείνουν ατιμόρυτοι οι άνθρωποι αυτοί. Αν θέλετε τις λεπτομέρειες, έχω το έγγραφο και φυσικά μετά την ακρόση αυτή μπορώ να σας το δώσω. ευχαριστώ. Και τώρα κανονικά θα πρέπει να πάρει ο κύριος Κασίδη το λόγο. Αλλά είχε κάποια προβλήματα στο ταξίδι του και έτσι δεν μπορούσε να φτάσει. Έχετε και γραπτό όμω την παρουσίασή του. Έχει μοιραστεί. Σας συνιστώ να τη διαβάσετε. Και έτσι πάμε. Είμαστε στο χώρο των διεθνών σχέσεων τον είδαμε, μας περιγράφει και τώρα πρέπει να δούμε τι σημαίνει η υλοποίηση της νομοθεσίας για τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και γι' αυτό θα δώσω το λόγο πρώτα στο Γενικό Διευθυντή της ΕΟΓΟΜΕΤΟΥ, τον κύριο Γκί Τιραν. Θα μας παρουσιάσει τις θέσεις της ε, Ένωσης στην οποία εκπροσωπεί. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τη γραμματεία της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου που μας έδωσε την ευκαιρία να μοιραστούμε κάποιες από τις ανησυχίες μας μαζί σας. Κάποια λόγια μόνο για να σας εξηγήσω τι είναι ακριβώς αυτή η Eurometo, ο χώρος που εκπροσωπώ εγώ, τον μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων έχει περίπου 500.000 κόσμο περιλαμβάνει βέβαια τα τρία τάφη χρυσό ταντάλο βολφράμιο, κασίτερο και χρυσό και προσπαθούμε να αναπτύξουμε μέσα στο πνεύμα της πράσινης οικονομίας, της ανάπτυξης στην Ευρώπη και εμείς τις προσπάθειές μας και μια συμπεριφορά στο μέλλον για μια ευρωπαϊκή κοινωνία η οποία χρειάζεται όλο και περισσότερα μέταλλα με τις ανανεώσιμες μορφές που έχουν αναπτυχθεί, με τα κλιματολογικά ισορροπημένα κτίρια, με το νέο σύστημα υγείας και όλα αυτά χρειάζονται αυτά τα μέταλλα. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να έχουμε ύψιστης ποιότητας επιδόσεις ε, περιβαλλοντικές, ενεργειακές, και ούτω καθεξής στην Ευρώπη. Για να συνεχίσουμε λοιπόν να το προσφέρουμε αυτό θα πρέπει να προσφέρουμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστική διάσταση της ευρωπαϊκής μας βιομηχανίας. Και... Με τον κανονισμό όσο έχει αυτή τη στιγμή παρέχονται ε, κάποιες ε, δυνατότητες ε, που αν δημιουργείται αυτή η αβεβαιότητα μπορεί να βλαφθεί η μη σιδηρούχα βιομηχανία στην Ευρώπη. Και το λέω αυτό συμμεριζόμενος απόλυτα το μέλημα να περάσουμε σε, μια, σε ένα αυξημένο πλαίσιο διαφάνειας όσον αφορά αυτά τα ορυκτά ε, που προέρχονται από ε, περιοχές ε, που έχουν εκραγεί ράξεις. Το να βρούμε λύσεις σε αυτό το πρόβλημα είναι προτεραιότητα για μας και στην ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέγεται ότι οποιαδήποτε σχέση με εμπόριο ευρωπαϊκής δράσης σε αυτόν τον τομέα πρέπει να τεθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της υλοποίησης της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και της ε, προοπτικής ε, συνεργασίας για την ανάπτυξη. Και θα πρέπει να δούμε το ε, κέλυφος αυτής της πολιτικής ε, και τις δραστηριότητε ε, για την ανάπτυξη. Είναι σημαντικό αυτά τα στοιχεία να μπορέσουν να ενταχθούν με πραγματιστικό ρεαλιστικό τρόπο ώστε η κατάσταση να διασφαλίσουμε ότι θα βελτιωθεί επί τόπου διότι αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα είναι αναγκαία για να βελτιωθεί η κατάσταση επιτόπου. Δεν χρειαζόμαστε, δεν θέλουμε ένα ε, επιβαρημένο γραφειοκρατικό σύστημα εκείνο που χρειαζόμαστε είναι η απάντηση στα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Από πλευρά βιομηχανίας ε, πλήρως δεσμευόμεθα για να υλοποιήσουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αυτό, επιτύχουμε αυτό το στόχο. Όχι μόνο σε σχέση με τα όσα προτείνονται από το νομοθέτημα Dodd Frank, που όπως αναφέρεται συνεισφέρει για να επιληθούν κάποια προβλήματα αλλά και διάφοροι άλλοι τομείς ε, του, των τριών τάφα και του χρυσού, κασιτέρου, βολφραμίου, ιτανταλίου και ε, του, του και ε, του χρυσού να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε ώστε σε μια εθελοντική ε, βάση να μπορέσουν να λειτουργήσουν προγράμματα ελέγχου και προτεραιότητες που δείχνουν ήδη επικερδή ε, ωφέλη σήμερα. Και στην πρωτοβουλία για την τροφοδότηση, αλυσίδα τροφοδότησης, ε, επίσης όσον αφορά την βιομηχανία παραγωγής, την ηλεκτρική βιομηχανία, πάλι για την τροφοδοσία της αγοράς, καθώς επίσης και η ε, Ένωση ε, Χρυσού καθώς επίσης ε, και η βιομηχανία Βολφραμίου. Όλα αυτά τα χιτήρια που αφορούν αυτά τα ορυκτά καλύπτονται από αυτή την πρωτοβουλία και θα, ακόμα και σε σχέση με τα χιτήρια όχι μόνο σε σχέση με την Ευρώπη αλλά και σε άλλες περιοχές. Τα χιτήρια στη ΗΠΑ για παράδειγμα στη Νότια Αμερική, στην Αυστραλία. Είναι ένα παγκοσμιοποιημένο παγκόσμιο σύστημα το οποίο υφίσταται και λειτουργεί με επιτυχία. Για να σας δώσω μόνο κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν την επιτυχία αυτή. Νομίζω το μέσο του Κασίτερου είναι ένα καλό παράδειγμα όπου από το 2010 μέχρι σήμερα 2014 έχουμε δραματικές αλλαγές όσον αφορά τους κανόνες τροφοδοσίας σε σχέση με προέλευση αυτού του μεταλλεύματος από την Αφρική για παράδειγμα το 2010 100% μπορείτε να δείτε ότι ήταν ε, η κάλυψη των αναγκών από την τροφοδοσία μας. Και με την ε, λειτουργία αυτού του εθελοντικού προγράμματος μειώσαμε αυτό τον όγκο. Υπήρξε λοιπόν αποτελεσματική δράση καθορίσαμε ποια ήταν ε, ε, τα μαύρα πρόβατα, οι ένοχοι, εκείνοι οι οποίοι θα έπρεπε να υποστούν κυρώσεις. Και σήμερα καταλήξαμε στα αποτελέσματα που έχουμε 99% σχεδόν δηλαδή 100% των των αναγκών μας ε, από πλευράς τροφοδοσίας ε, είναι ε, προέλευσης καθαρής. Όχι μόνο ευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εδραστούμε και να αναπτύξουμε τα ωφέλη αυτού του συστήματος και να πούμε ότι από κοινού με το νομοθέτημα Dodd-Frank αυτά τα συστήματα όχι μόνο συνδέονται με το εμπόριο αλλά συμπεριλαμβάνουν και κίνητρα για να εμπλέκεται όλη η αλυσίδα δημιουργίας ε, πρόσθετης αξίας ε, καθώς επίσης και την ανάπτυξη αναπτυξιακών προγραμμάτων και όλα αυτά καταδεικνύουν επιτόπου χειροπιαστά ωφέλη τα οποία συνεπάγονται. Είμαστε λοιπόν μια βιομηχανία παγκόσμιας ε, εμβέλειας. Ε, το να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη σε αυτές τις δραστηριότητες είναι κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της βιομηχανίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό όμως χωρίς να λάβουμε υπόψη ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μία από αυτές τις ανάγκες είναι η ανάγκη να υπάρχει ένα ισοδίκαιο, ισότιμο πεδίο εφαρμογής και δραστηριοποίησης παγκοσμιοποιημένα. Το να επιληθούν τα προβλήματα μόνο στις, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη ΣΥΠΑ με το νομοθέτημα για παράδειγμα Dodd Frank θα έχει μόνο περιθωριακή επίπτωση. Και από αναλύσεις που έχουν γίνει σε σχέση με αυτές τις προτάσεις ε, βλέπουμε ότι μόνο 5%, 5 των χιτηρίων παγκόσμια έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη. <coughs> Μία τέτοια προσέγγιση λοιπόν θα είχε μόνο αποτέλεσμα στο 5% των ε, προβλημάτων. Πέρα από όλα αυτά πρέπει είναι ανάγκη να εξετάσουμε ότι αν δεν αναπτυχθεί η αλυσίδα τροφοδότησης και αν δεν υπάρξουν κίνητρα για να διαμορφωθεί και να προσαρμοστεί με τις, ανάλογα με τις ανάγκες αυτή η αλυσίδα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να αγοράζουν από μη καθαρές πηγές από την Κίνα ή από οπουδήποτε αυτά τα ορυκτά όπου θα συνεχίσουν μη πιστοποιημένες δράσεις χωρίς διαπίστευση να ε, οδηγούν στην εξ εξόριξη αυτών των ορυκτών και στην εισαγωγή τους. Το να δημιουργήσουμε λοιπόν μια μεγαλύτερη τέτοια εξάρτηση από τρίτες χώρες θα είναι μια συνέπεια, θα είναι μικρότερη πρόσθετη αξία που θα παράγεται σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποτύχουμε να διασφαλίσουμε τις ανάγκες μας από την τροφοδοτική αλυσίδα για τα συγκεκριμένα ορυκτά, υπονομεύοντας τους στόχους της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση επιτόπου. Έχουμε μια σειρά συστάσεων που αναπτύχθηκαν και εκπονήθηκαν και σε σχέση και με τις ε, αρμόδιες ε, γαλλικές αρχές. Ε, αφορούν την απουσία σαφήνειας και βεβαιότητα στο σύστημα. Το πώς θα αναπτυχθεί το σύστημα έχει σήμερα κάποιες, συνεπάγεται κάποιες αβεβαιότητες δεν υπάρχουν πλέον κίνητρα για να επενδύσει κανείς στην Ευρώπη. Και το κύριο στοιχείο στο να βελτιωθεί η σαφήνεια ε, αυτού του συστήματος είναι για μας κύρια προτεραιότητα. Απαριθμό και άλλες ανησυχίες και μελήματα το να ε, υπάρξει δυνατότητα να ε, εξαιρεθούν ε, κάποιοι τομείς και το να μπορέσουμε να συμμεριστούμε και να εμπλακούμε πλήρως με τις αρχές που θα προτείνει ένα ευρωπαϊκό σύστημα για να συμμορφωθούμε με τον κανονισμό. Ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση με το ενισχύει σύστημα συμπεριλαμβάνοντας και τις ε, οδηγίες ε, του ΟΣΑ για την δέουσα ε, επιμέλεια καθώς επίσης και τα στοιχεία Ντόντ Frank. Επίσης υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο συνδέεται με το ισοδίκαιο πλαίσιο δραστηριοποίησης στην ενιαία εσωτερική αγορά. Ένας τρόπος να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και να μην υπάρξει κακοφωνία και κατακερματισμένος ε, ε, κατακαιρματισμένη υλοποίηση είναι να δημιουργηθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή αρχή που θα ελέγχει τη συμμόρφωση με αυτόν τον κανονισμό και θα ε, παρέχει περαιτέρω από ε, σαφήνεια μέσω ελέγχων τρίτων ε, μερών και θα υπάρχει δυνατότητα διασφάλισης του απορρίτου των στοιχείων. Με αυτά μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσεις είτε σε εμένα είτε στους συναδέλφους που είναι παρόντες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις στην παρουσία σας και τις συμβουλές που ε, μας δώσατε. Επόμενος αγορητής ε, είναι ο κύριος Τζούλιαν Λάγκαρτ. από την Digital Europe, μέλος του, του ομίλου ε, ορυκτών μεταλλευμάτων από περιοχές ε, συγκρούσεως. Έχετε το λόγο. Mr. Chairman, um... Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, κύριε και κύριοι, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σήμερα. Εργάζομαι και την Intel. Ταυτόχρονα εκπροσωπώ την ε, Digital Europe, τον ευρωπαϊκό κλάδο δηλαδή της ψηφιακής τεχνολογίας. Πρόκειται για ένα σημαντικό κλάδο που αποτελεί και τη ρεχοκοκαλιά της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, οικονομίας, κοινωνίας που τόσο μεγάλη σημασία αποδίδει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι για μας προτεραιότητα, ακούσαμε ήδη αρκετά για τα περίφημα τρία ταφ και το, χριστό και το χρυσό, ταντάλιο, βολφράμιο, κασίτερο και χρυσός που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά, ιδιαίτερα δε το βολφράμιο και ο κασίτερος. Έχουμε από την αρχή τηρήσει τις ε, προδιαγραφές. Η Έριξον και η Philips έχουν ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές να τηρούν. Πολλά ακόμα μένουν να γίνουν βεβαίω χωρίς να είναι βέλτιστα τα αποτελέσματα πάντοτε. Θα ήθελα να, εκφράσω, να εξηγήσω τι έχουμε κάνει εμείς και πώς έχουμε εμείς συμβάλει στο, στο διάλογο αυτόν. Απλώς δεν είμαστε όμως ένας τομέας που απλώς καταναλώνει αυτά τα μεταλλεύματα για να είναι αποτελεσματικός ένας κλάδος. Θα πρέπει να κινούνται όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια συντονισμένη προσπάθεια. Είμαστε ένας κλάδος που δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει μια, διευρύ, ε, μια ευρεία αλυσίδα προμηθειών σε διάφορα επίπεδα, άνω των 7 επίπεδων, χιλιάδες στοιχεία και επιχειρήσεις μετά το δεύτερο επίπεδο. Όμως, στις προμήθειες δεν έχουμε καμία κανέναν έλεγχο ως προς την αλυσίδα της προμήθειας, με το δεύτερο επίπεδο προμήθειας. Κάνουμε λοιπόν έναν διάλογο με εμπλοκή όλων των εμπλεκομένων για να έχουμε στο δυνατόν πιο υπεύθυνη συμπεριφορά και εμπόριο ακόμη και στις περιοχές ψηλού κινδύνου. Υπάρχουν ε, πολλές φορές επίπεδα άνω των 7 στην παραγωγή από το ανώτερο μέχρι το κατώτερο επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής και θέλουμε να επικεντρωθούμε κυρίως στα χιτήρια και τις μονάδες τήξεως. Έχουμε εδώ έναν σχετικά πιο περιορισμένο αριθμό παραγόντων από την είναι τα ορυχεία παραδείγματα και αποτελούν και ασφαλή τρόπο να ε, ελεγχθούν, να επιβεβαιωθεί η αλυσίδα και η προέλευση. Ενώ δεν είναι το ίδιο πράγμα δυνατό για τα ε, ορυχεία. Το πρόγραμμα CFS που συμπεριλαμβάνει και άλλους τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, αεροβιομηχανία έχει βοηθήσει ιδιαίτερα στη βελτίωση της κατάστασης στην ε, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και την αποφυγή των ε, δραστηριοτήτων των επιχειρηματικών στην περιοχή όταν υπάρχουν ε, προβλήματα όπως συγκρούσεις κτλ. Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο, το CFS, το οποίο ε, βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό επικαιροποίηση, υπό ενημέρωση για να καλύψει και νέους τομείς. Θα πρέπει, πιστεύουμε, να ασκείται από τον καταναλωτή η πίεση κατά του χιτηρίου ή του, της μονάδας τήξεως και εξευγενισμού, διότι εκεί ακριβώς θα αισθανθούν την πίεση. Άρα λοιπόν μετά το βήμα αυτό της ε, τήξης είναι πια δύσκολο να διαγνωστεί εάν προέρχεται από περιοχή συγκρούσεων το μετάλλευμα ή όχι. Το σημείο τήξη είναι και το τελευταίο σημείο στο οποίο μπορεί να διαγνωστεί το πρόβλημα αυτό και γι' αυτό θέλουμε να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία η οποία είναι και συμπληρωματική σε σχέση με το νόμο Dodd Frank των Πολιτειών. Πιστεύουμε ότι κίνητρα για την ε, λειτουργία του συστήματος αυτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορούν να επαρκέσουν στο πλαίσιο των εφιστομένων μέσων όπως δηλαδή το τμήμα 1502 του νόμου Ντότ Φρανκ, οι κατευθυντήριες γραμμέ του ΩΣΑ που εξετάθησαν νωρίτερα, οι εθελοντικές πρωτοβουλίες που ήδη λειτουργούν και ασκούν σημαντική πίεση στην αγορά. Ε, αν όμω καταστεί υποχρεωτικό ο κανονισμός, ενδέχεται να οδηγήσει σε ακόμη πιο πολλές δυσκολίε για τα χιτήρια και τις μονάδε επεξεργασία ω προ την ε, τήρηση των όρων του και να οδηγήσει σε ακόμη περισσότερα προβλήματα γενικά. Έτσι λοιπόν, το πρότυπο για την ε, έκθεση και λογοδοσία που ονομάζεται IPC 1755 διευκολύνει την επικοινωνία στην αλυσίδα προμήθειας και μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση της πορείας ενός μεταλλεύματος, ενώ πιο αυστηρές διατάξεις θα μπορούσαν να είναι υπερβολικά επιβαρυντικές. Ασφαλώς πρέπει να υπάρξει μια γενική προσέγγιση, μια παγκόσμια προσέγγιση και έλεγχος διεθνής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί και πρέπει να διαχειριστεί το λευκό ή ανοιχτό κατάλογο χιτηρίων, δηλαδή των μη, αποκλει... των μη αποκλεισμένων χιτηρίων, μαζί με τον ΩΣΑ και το θέμα της δέουσας προσοχής με το βήμα υπαριθμών 5 των κατευθυντηριών γραμμών του ΩΣΑ μπορεί να συμβάλλει στην αποκάλυψη των μη χρηματοοικονομικών ε, πληροφοριών με τις οποίες μπορούν οι επιχειρήσεις να δείξουν περισσότερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη διαθέση των πληροφοριών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις αντίστοιχες με αυτές των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Όταν καλούνται να δώσουν στοιχεία για, τα, ε, για την πρόληψη των προϊόντων τους ή να λογοδοτήσουν για την αλυσίδα τη προμήθεια. της προμήθειας. Είναι πιο δύσκολο όμως αυτό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν έχουν πόρους, δεν έχουν προσωπικό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν περιορισμένο δε δυναμικό διαπραγματευτικό σε σχέση με τους μεγαλύτερους πελάτες ή προμηθευτές. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι δύσκολο για μια μικρομεσαία επιχειρήση να εξασφαλίσει τις πληροφορίες από τον μεγάλο προμηθευτή της για την αλυσίδα ενώ μεγαλύτερες επιχειρήσεις, μεγαλύτερη δύναμη στην αγορά θα το κατάφερναν. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς την υλοποίηση αυτών των όρων για τις προμήθειες, γιατί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτό μπορεί να συνεπάγεται και de facto αποκλεισμό από την ε, αγορά των δημοσίων ε, διαγωνισμών. Το κόσμο επίση η χρηματοδότηση κόσμου μπορεί να, θα πρέπει να διατεθεί για όλες τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν καλούνται να εφαρμόσουν τι κατευθυντήριες γραμμές του ΩΣΑ, ανεξαρτήτω του αν εισάγουν τα καλε, τους τις καλυπτόμενες πρώτες ή αν βρίσκονται σε περαιτέρω στάδιο της αλυσίδας της προμήθειας. Είναι σημαντικό επίσης να οικοδομήσουμε πάνω σε φυστάμενα σχήματα, όπως είναι το CFSP, όπως είναι οι υπεύθυνε προδιαγραφές χρυσού, όπως είναι η αλυσίδα πιστοποίησης και παρακολούθησης στον τομέα των κοσματοπολών, όπως είναι η πρωτοβουλία τη ICMC για το βολφράμιο. Πρέπει να πούμε ότι πρέπει να προσδιοριστεί τι σημαίνει ακριβώς ε, περιοχή πληττόμενη από σύγκρουση και περιοχή υψηλού κινδύνου. Πρέπει να μην στιγματίζονται βεβαίω οι περιοχέ, αλλά πρέπει και ταυτόχρονα μια επιχείρηση να μπορεί να καταλάβει, να εντοπίσει αμέσω ποια είναι αυτή η περιοχή που παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο ή είναι πλήττονται από σύγκρουσες. Ε, και εκεί θα πρέπει να γίνεται η ειναι υπλητα απο συγκρουσει και αντιστοιχα εκει θα πρεπει να γινεται η προσπαθεια για την ανάπτυξη του δυναμικού, για τη βελτίωση των υποδομών. Όλα αυτά χρειάζονται πολύ χρόνο. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, υποστηρίζουμε τις προτάσει τη Ευρωπαϊκής Ένωση, στηρίζοντας τις προτεγραφέ του οργανισμού του ΟΟΣΑ με την δέουσα προσοχή για τις επιχειρήσεις, που σημαίνει περιορισμό του κίνδυνου, όχι εκμηδενισμό. συμπληρώνει το, την παράγραφο 1502 του νόμου Dodd-Frank. Τίνει να ελέγξει στο πρώτερο επίπεδο των προμηθειών με, ευρύτερο γεωγραφικό, με ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη το πρόβλημα. Προσφέρει ένα πακέτο που περιλαμβάνει και συνοδευτικά μέτρα και συνομιλεί με τις εμπλεκόμενες χώρες. Και πιστεύουμε ότι χρειάζεται κατεπηγόντως να αναπτυχθεί ο τεχνικός διάλογος σε πολυμερές επίπεδο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Είναι περίπλοκα τα πράγματα, επικρατεί αρκετή σύγχυση, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε και τι δυνατότητες υπάρχουν και πώς μπορεί ένας νέος μηχανισμός, ένα νέο σύστημα να προσφέρει θεμένη αξία. Θα θέλαμε λοιπόν να αναπτυχθεί ένας πολυπλευρός διάλογος με όλους τους εμπλεκομένους. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, τελευταίος τώρα ο κύριος Μάικλ Γκίμπ επικεφαλής εκστρατείας για τους σπόρους που προέρχονται από περιοχές πληττόμενες από συγκρούσεις. Ευχαριστώ. Η Global Witness ε, έχει έρευνα το σχέση μεταξύ του εμπορίου ε, στα ορεικτά και της παραβίασης ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εργαζόμαστε για χρόνια και χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και ευχαριστούμε που μας καλέσατε σε αυτή τη σημαντική συζήτηση. Εδώ δεν εκπρόσωπο μόνο την Global Witness, αλλά εκπροσωπώ και τον συνασπισμό της κοινωνίας των πολιτών που ε, εκπροσωπεί πάνω από 60 οργανώσεις κοινωνίας πολιτών όπως η Διεθνής Αμνηστία και άλλες οργανώσεις παρά το γεωγραφικό εύρος ε, της δουλειά μας από την Κολομβία μέχρι την Κεντρική Αφρική και τη Ζιμπάμπουε και τη Μιαμάρ. Ε, το θέμα της ε, επίλυσης των συγκρούσεων είναι ένα θέμα που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό και οδηγεί σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλοι θέλουμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Σήμερα θα ξεκινήσω από το εξή. Όλοι όσοι έχουν περάσει χρόνο σε αυτές τις κοινότητες ε, από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσει οποιοδήποτε. Η σημερινή κατάσταση δεν είναι πολιτικά βιώσιμη, ούτε οικονομικά βιώσιμη, ούτε μπορούμε να την περισπεστούμε ηθικά. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Ήδη ακούσαμε τα αποτελέσματα αυτού του εμπορίου σε ορισμένα τμήματα του Ανατολικού Κογκό όπου χρηματοδοτούνται ομάδες ε, που προβαίνουν σε σεξουαλικά εγκλήματα, σε εκτοπισμούς και σε δολοφονίες. Όμως ε, το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Μέσα σε λίγες μέρες θα έχουμε τη δεύτερη επέτειο της ε, πρόσφατης σύραξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Εδώ μιλάμε για μια χώρα που το 1 τέταρτο του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί από το σπίτι του και το 50% του πληθυσμού χρειάζεται επιγόντως ανθρωπιστική βοήθεια. Σύμφωνα με μια έκθεση πρόσφατη που έγινε από τη Global Witness, εμπόριο σε χρυσό, διαμάντια, ελεφαντόδοτο και ξυλία χρηματοδοτούν και τις δύο πλευρές αυτής της σύραξης ε, και ε, φυσικά αποστορπείται περισσότερο η κατάσταση. Περίπου δύο τόνοι χρυσού ε, κάθε χρόνο μπαίνουν παράνομα, βγαίνουν παράνομα από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στο βόρειο τμήμα της χώρας ε, υπολογίζεται ότι ε, κερδίζουν ε, αυτές οι ομάδες 120.000 ευρώ το χρόνο και περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ έχουν βγει από τη χώρα από τότε που αναστέλει βγήκε η χώρα από τη διαδικασία Κίμπερ Φυσικά εδώ τέτοιε σειράξει δεν μπορούν να σταματηθούν αν δεν υπάρχουν σοβαρές προσπάθειες για να καταπολεμηθεί αυτό το εμπόριο που είναι τόσο κερδοφόρο. Κάτι πρέπει να αλλάξει και χαίρομαι που ακούω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση την ιδέα ότι ε, μεγάλα κέντρα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι μέρος της λύσης. Είναι αναμφισβήτητο ότι ε, υπάρχει μια παγκόσμια εταιρική ευθύνη για να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις δεν θα συνεισφέρουν ε, στην κατάχρηση και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αρχές, κατευθυντήριες αρχές το 2011 των ΗΠΑ το καθιστούν αυτό και εδώ πιστεύουμε ότι επισέρχεται ιδέως επιμέλεια από το 2010 όλες οι εταιρείες που μπορεύονται φυσικούς πόρους μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τον οδηγό δέσους επιμέλειας του ΟΣΑ που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη βιομηχανία και τι επιχειρήσει. φυσικά. Πρέπει να είμαστε σκεπτικοί για μεγάλε ιδέε που επιτίθεται ότι θα λύσουν πολύπλοκα προβλήματα, αλλά ιδέω επιμελή δεν είναι μια μεγάλη λύση αυτό που ενθαρρύνει ιδέω επιμέλεια στην πράξη είναι οι τοπικέ κοινότητε, οι εταιρείε, οι τοπικέ κυβερνήσει, αυτοί ε, που λειτουργούν σε αυτά τα περιβάλλοντα να συνεργαστούν για να εντοπίσουν ε, του κινδύνου που του απειλούν ε, και αντίθετα με αυτό που μπορεί να, και να δρουν τι μπορεί να γίνει για να μετριαστούν οι κίνδυνοι αυτοί στι κοινότητέ του. Ιδίω η επιμέλεια είναι μια διαδικασία ευέλικτη, δεν είναι γραφειοκρατική διαδικασία Πολλές ε, εταιρείε κάνουν κάποια πράγματα στα δικά τους ε, περιβάλλοντα και μιλάμε για ένα νέο τρόπο του να κάνει κάποιος ε, επιχειρήσεις και να έρχεται σε επαφή με τις κοινότητες αυτές που προσφέρουν αυτούς τους πόρους Επίσης Πιστεύουμε ότι πρέπει να ενδυναμωθεί η σημερινή πρόταση. Για πολλές εταιρείες, ιδέω επιμέλεια, είναι πραγματικότητα. Ήδη η αλυσίδη εφοδιασμού ε, εφαρμόζει τέτοιες υποχρεωτικές απαιτήσει όπως στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, μόνο 7 με 12% των εταιριών που δεν θίγονται απευθεία από τον νόμο Dodd ε, Frank έχουν ξεκαθαρίσει ότι η έχουν τέτοιες ε, πολιτικές διαθέσιμες ε, εμείς πιστεύουμε ότι η εταιρεία επιμέλεια θα αλλάξει τη συμπεριφορά των εταιριών. Αν γίνει υποχρεωτικό αυτό το σύστημα θα είμαστε σίγουροι ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείε λειτουργούν βιώσιμα και με διαφάνεια. Θα μιλήσουμε με μία ενιαία φωνή όταν θα προσπαθήσουμε να αποφθυνθούμε στα χιτήρια και στι εγκαταστάσεις τήξης, ακόμη και σε αυτούς που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε διαθέσιμες πληροφορίες και φυσικά θα πρέπει ε, να καταστήσουμε πιο εύκολο τις εταιρείες ε, να ε, δραστηριοποιούνται πιο υπεύθυνα σε περιοχές με σειράξεις όπου χρειάζονται περισσότερο τέτοιες επενδύσεις. Καταρχήν θα πρέπει να κινηθούμε προς τους κανόνες της δέουσας επιμέλειας και ίσως θα πρέπει να δούμε πώς θα ακολουθήσουμε και τις υφιστάμενες, ε, την υφιστάμενη νομοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, θα καλύπτονται όλα, ε, όλες οι ύλες που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξάρτητα με τον τρόπο και τη μορφή τους αλλά φυσικά πρέπει να λάβει κανεί υπόψη το πολύ μεγάλο αριθμό μικρών και μεσών επιχειρήσεων Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλέ διαδραματίζουν ε, ένα σημαντικό ρόλο στον, ε, στο εμπόριο αυτών ε, των μετάλλων, κυρίω του χρυσού. Φυσικά πολλοί έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν να θεωρούνται εταιρείε δεύτερη κατηγορία και να είναι εκτό τη νομοθεσία. Πρέπει να θυμόμαστε ότι πολλές ευρωπαϊκές ΜΜΕ φύγονται ήδη από ε, νομοθεσία δέουσας επιμέλειας. Ε, για αυτές τις εταιρείε είναι ήδη πραγματικότητα η δέουση επιμέλεια και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα αυτές τις επιχειρήσεις. Καθώς ε, είπαμε, ο οδηγός δέουσας επιμέλειας του ΩΣΑ είναι ευέλικτος ήδη ρυθμίζει το είναι θέση της εταιρείας στην αλυσίδα του εφοδιασμού ε, πρέπει να γίνουν κάποιες κατάλληλες προσπάθειες. Ε, μιλά για τη ροή των πληροφοριών που εξελίσσεται με το χρόνο. Επίσης, ε, δίνει έμφαση στο να συνεργαστούν οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις μέσω διάφορων προγραμμάτων. Νομίζουμε ότι αυτό πρέπει να ενθαρρύνουμε, εξομαλύνοντας τη διαδικασία της δόσης επιμέλειας και δημιουργώντας μια συλλογική ζήτηση, έτσι ώστε όλες οι εταιρείε να μπορούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις και με το αίτημα των πελατών τους. Θα πω αυτά που είπα νωρίτερα, κάτι πρέπει να αλλάξει. Φυσικά είναι ζωτικό να διασφαλίσουμε ότι η αλλαγή που θα φέρουμε θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Καλωσορίζουμε το γεγονός ότι η πρόταση της Κομισιόν έχει ευρία γεωγραφική εφαρμογή και δεν απομονώνει μία συγκεκριμένη περιοχή έτσι ώστε να δημιουργηθούν στρεβλώσει στην αγορά και επίσης καλωσορίζουμε κάποια συνοδευτικά μέτρα που ακούσαμε από την ανακοίνωση που θα διασφαλίσουν ότι αυτός ο κανονισμός θα συνοδεύεται από πολιτικές που ε, θα καταπολεμούν ε, τις παρενέργειες. Όμως ε, πιστεύουμε ότι η συζήτηση θα πρέπει να γίνει παράλληλα με τη συζήτηση για τον κανονισμό. Έχουν υπάρξει κάποιε συζητήσει για τον αντίκτυπο του νόμου Dodd Frank. Δεν έχω χρόνο για να αναφερθώ σε αυτό λεπτομερό, αλλά θέλω να πω ότι στα 10 χρόνια που η Global Witness εργάζεται σε αυτό το θέμα ποτέ δεν είδαμε τόσο μεγάλη αλλαγή επιτόπου όπω αυτή που έγινε κατόπιν ε, τη ε, εφαρμογή τη υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια στην ΕΠΑ. Έχουν αλλάξει το πώ λειτουργούν οι τοπικοί φορείς και ανταλλάσσουν πληροφορίε και έχουν δημιουργηθεί πολύ μεγάλε δραστηριότητες. Ε, επίσης, έχει δοθεί προσοχή στις συνθήκες εργασίας των εργατών, κυρίως μικρής κλίμακας και ε, Επίσης, ε, πολύ νωρίς ξεκινά η διαδικασία και μειώνεται η εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων από αυτές τις ενόπλες ομάδες. Πιστεύουμε ότι η δέωση επιμέλεια παρέχει την ευελιξία και την απάντηση που χρειάζεται και πιστεύουμε ότι, ότι χρειαζόμαστε περισσότεροι και όχι λιγότεροι από αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα οι ευρωβουλευτές, τα μέλη που ζήτησαν να παρέμβουν. Ο Χέλμουτ ήταν ο πρώτος. Αρένα, Γιούντιτ. you have and Ms. and Emma. Okay, Helmut. Λοιπόν ο Χέλμουτ πρώτος, παρακαλώ. Ευχαριστώ Μπέρντ. Ευχαριστώ τους πραγματογνώμονες για τις παρεμβάσεις και εισηγήσεις τους. Κατέστησαν σαφές ότι εδώ πρόκειται για ένα πολύ περίπλοκο σύνθετο θέμα και είναι επιτέλους η χρονική στιγμή ως συγκυρία να ρυθμίσουμε τις διατάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις. Και με την παρουσίαση στο διαδίκτυο όλων αυτών ελπίζω ότι ιδιαίτερα η παρέμβαση του κυρίου ε, θα βρει την σωστή απήχηση. Θα πρέπει ως ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή να δράσουμε ώστε η, επιθυμή, η ε, συνεισφορά αυτών των ε, τομέων να μπορέσουν να, η συνεισφορά να μπορέσει να τονιστεί και θετικό είναι το ότι από αυτή την παρέμβαση απορρέουν δυνατότητες στα προβλήματα να τα φωτίσουμε και να δούμε πώς πρέπει να κινηθούμε. Αυτά τα οποία είχαμε συζητήσει σύντομα κατά το παρελθόν, ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των δεσμεύσεων αυτών και των ρυθμίσεων από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή και να ολοκληρωθεί. Και όπως εκφράστηκε και εξάλλου και στην ακρόαση, σαφέστατα πρέπει να διευρυνθεί η προσέγγιση αυτή όσον αφορά τις γεωγραφικές ε, ε, περιοχές ε, και όσον αφορά τα, τις αρχές προέλευσης. Ενδιαφέρουσα ήταν η παρέμβαση σε σχέση με τον ΩΣΑ, να σκεφτούμε σε σχέση με τις προτάσεις του ΩΣΑ. Μήπως η συνολική αλυσίδα τροφοδοσίας ανεξάρτητα από την έδρα επιχείρησης επεξεργασίας να λαμβάνεται υπόψη και οι κατευθυντήριες γραμμές του ΩΣΑ στην ελαστικότητά τους να είναι ο μύτος της Αριάδνης με τον οποίο θα κατευθυνθεί και θα δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να δώσω τη δυνατότητα σε όλους τους, δυνατό, σε όλους τους συναδέλφους να παρέμβουν και δεν θέλω να περιορίσω το χρόνο τους μακρηγορώντας. Σε σχέση με τον ε, εκπρόσωπο που μίλησε προηγούμενα, ε, είπε ότι είναι υπέρ αυτής της ρύθμισης. Δεν είπε όμως αν η ε, εθελούσια δέσμευση είναι επαρκής ή αν θα πρέπει να υπάρχει μια οικουμενική ρύθμιση ίση και ίδια για όλους όσον αφορά την πρόσβαση ε, ε, στην αγορά που θα δέσμευε όλους μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο. Και θα πρέπει αυτό και στις διμερείς ε, συμφωνίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλα κράτη να βρει την απήχησή του. Ένα σημείο που για την TTIP, ε, τη Συμφωνία Επενδύσεων και Εμπορίου με τις ΗΠΑ, θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μπορούσε να τύχει συνέχεια και ίσως να ενταχθεί και αυτό. Και εξάλλου επίσης μέσα στο πλαίσιο του ΠΟΕ, αν θα έπρεπε να εκφράσουμε σαφέστερα ότι μόνο δεσμευτικού χαρακτήρα ρυθμίσεις και διατάξεις θα πρέπει να εντάσσονται που με σαφή τρόπο θα μπορούν να ελέγχονται, να επιτηρούνται και να αποβαίνουν προς όφελος ε, των ε, πολιτών ε, ιδιαίτερα όταν έχουμε προβλήματα περιοχών σε σύραξη. Ευχαριστώ. Αν έχετε μια συγκεκριμένη ερώτηση σε κάποιον από τους επαΐοντες θα βοηθούσε. Συγκεκριμένη ερώτηση λοιπόν και έτσι να συνεχίσουμε. Η Μαρία παρακαλώ. Merci. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμονες με τις εκθέσεις τους που επιτρέπουν έτσι να διευκρινιστούν οι θέσεις των μεν και των δε. Ε, θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στο γενικότερο ρόλο που έχουμε να επιτελέσουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν μιλούμε για ε, συγκρούσεις συχνά ε, σπρώχνουμε τις ευθύνες στο επίπεδο της τοπικής διακυβέρνησης. Εγώ νομίζω όμως ότι τώρα πρέπει να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να μην μεταθέτουμε τις ευθύνες στην τοπική διακυβέρνηση και γιατί όντω πολλές φορές για τις ευθύνες λέμε «Α, μπορεί να φταίει είτε η τοπική διακυβέρνηση είτε ο ίδιος ο καταναλωτής» γιατί έχει την επιλογή όταν πρόκειται να καταναλώσει κάτι θα πρέπει να επιλέγει την, ε, ε, το δίκαιο εμπόριο, αυτό που σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, και τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Αυτό έχει επιλέξει η Επιτροπή με την εθελοντική προσέγγιση, δηλαδή ε, να παίξει η αγορά το ρόλο της επιλογής. Όταν μια επιχείρηση δεν τηρεί τους κανόνες θα πρέπει να προσαρμόσεται η αγορά, δηλαδή ο καταναλωτής. Και να πει αν δεν τηρεί αυτή η επιχείρηση τους κανόνες του παιχνιδιού δεν θα πάω να αγοράσω από αυτή την επιχείρηση. Ναι, αυτό συνεπάγεται ότι δείχνουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην αγορά για αν δούμε ποιε είναι οι εθελοντικέ προσεγγίσεις αυτή τη στιγμή, αποδεικνύεται ότι η αγορά δεν φέρνει τόσο γρήγορα αποτελέσματα ή τόσο εύκολα αποτελέσματα. Παίρνει μη τι άλλο πολύ χρόνο για να αποδώσει ο έλεγχος αγοράς. Και εδώ δεν μιλώ για ανταγωνιστικότητα. Και σε αυτό απευθύνομαι προς του εκπροσώπους των επιχειρήσεων. Μιλούμε για ε, ανθρωπινε ζωέ. Αν λοιπόν συγκρίνουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη βάλουμε στην πλάστιγκα μαζί με τις ανθρώπινες ζωές που κινδυνεύουν στις χώρες όπου, που πλήττονται από συγκρούσεις, εγώ νομίζω ότι θα έχω εύκολη επιλογή. Γιατί ναι, θέλω να υποστηρίξω την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Αλλά εάν και βλέπουμε τον, τον Global Business που ήρθε να μας μιλήσει για τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται στην περιοχή του Κιβού, του Κιβού στο Κονγκό, αλλά όχι μόνο στο Κιβού, αλλά και αλλού. Ευθύνη μας είναι λοιπόν να λάβουμε μέτρα που δεν είναι μέτρα αγοράς, αλλά μέτρα υποχρεωτικά. Συγκεκριμένη λοιπόν ερώτηση. Λέγεται καταρχάς ότι η εθελοντική αυτή ε, προσέγγιση φέρνει αποτελέσματα και μάλιστα εκπρόσωπος από την Ρομετό μας λέει ότι για τον Κασίτερο έχει φέρει 100% αποτελέσματα και ότι η αλυσίδα του Καστέρου είναι 100% καθαρή. Ποιος μας το λέει όμως ότι είναι καθαρή, η αυτοπίστωση, η αυτοπιστοποίηση, το κάνει αυτό ο ίδιος ο κλάδος του Καστέρου. Και αν πάει τόσο καλά, δεύτερη ερώτηση, γιατί να μην είναι υποχρεωτικό, αφού μπόρεσε δηλαδή τόσο εύκολα να εφαρμόσει τους κανόνες, δεν αποδεικνύεται ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια φάση που πρέπει να προωθήσουμε το θεμητό ανταγωνισμό, δηλαδή να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες ακολουθούν την καθαρή αλυσίδα προμήθειας για να μην ενισχυθεί ο αθέμητος ανταγωνισμός από εκείνες που δεν την ακολουθούν. Άρα πρέπει να επιλέξουμε την υποχρεωτική προσέγγιση. Επίσης, είναι μόνο 5% εκείνα τα χιτήρια τα οποία δεν καλύπτονται. Ναι, έστω. Να μην μιλούμε μόνο για χιτήρια, να φτάνουμε μέχρι το τελικό προϊόν όμως, εάν θέλουμε μια ουσιαστική αποτελεσματικότητα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί δεν πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τελικό προϊόν. Και θα σώσω το παράδειγμα της γεωργικής παραγωγής για τρόφιμα που ξέρετε ότι ήμασταν πολύ προσεκτικοί και θέλουμε ο Ευρωπαίος καταναλωτής να έχει στο πιάτο του προϊόντα που εγγυώνται την προστασία του. Αναπτύχθηκαν λοιπόν στον κλάδο αυτών της γεωργίας τροφίμων μηχανισμοί που μπορούν να εγγυηθούν την ίχνη λασιμότητα από το πρώτο στο τελευταίο στάδιο. Γιατί λοιπόν αντίστοιχοι μηχανισμοί δεν μπορούν να θεσπιστούν στους τομείς που μας ενδιαφέρουν σήμερα, τα μέτρα δηλαδή και την κατεργασία τους μέχρι τον τελικό χρήστη, ώστε ο τελικός χρήστης, ο Ευρωπαίος καταναλωτής, να ξέρει ότι χρησιμοποιώντας τα δεν συμβάλλει στους θανάτους και τους φόνους αθώων στις χώρες από, την οποία, από τις οποίες τα μεταλλεύματα. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να έχουμε την ίχνη λασιμότητα για λόγους ανθρωπιάς και ανθρωπισμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Judith. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό ε, είναι ένας κανονισμός που έχει ένα αναπτυξιακό σκοπιό, ένα σκοπό να σπάσουμε αυτή την κατάρα των πόρων και έχει και το στόχο να υπάρχει βιώσιμη μεταλλευτική δραστηριότητα σε τέτοιες δύσκολες περιοχές. Η κύρια μου ερώτηση είναι, αν δούμε την πρόταση που έχουμε επιτάπητος, δημιουργούμε πράγματι ζήτηση στην Ευρώπη για αυτά τα ορυκτά που τα παίρνουμε από τέτοιες ασταθείς περιοχές ή περιοχές με σειράξεις. Και νομίζω ότι κάποιος πολύ κλαφυρά το είπε προηγουμένως. Αν αυτή είναι μια πολιτική που δεν ζημιώνει, τότε τελικά δεν κάνουμε και τίποτα καλό. Και νομίζω ότι έχουμε τρία επίπεδα λήψη αποφάσεων. Ε, θα έχουμε υποχρεωτικό χαρακτήρα ή εκούσιο. Θα, ακολουθεί, θα, θα καλύψουμε εκεί και τα καρλωτικά αγκαθά ή μόνο τις πρώτες Και επίσης ε, θα ε, προσπαθούμε να επικεντρώσουμε τα πάντα στα χιτήρια και σε εγκαταστάσεις τήξης και στην Νοτιοανατολική Ασία. Θα πάμε κατάντι, δηλαδή θα πάμε ανάντι μέχρι το ορυχείο με τις δραστηριότητε αυτές. Επίσης, η ερώτησή μου έχει να κάνει, μάλλον απευθύνεται στον Διευθυντή της Ρωμετό που είπε ότι δεν υπάρχουν κίνητρα για τα χιτήρια και τις εγκαταστάσεις τήξης να κάνουν το σωστό. Αυτή είναι μια ερώτηση που θέλω να του θέσω. Ποια κίνητρα εσείς θα αναζητούσετε προκειμένου τα χιτήρια που δεν είναι σε ευρωπαϊκό έδαφος να, ε, να συνεχίσουν να μάλλον ε, αυτά τα χιτήρια να συνεχίσουν να παίρνουν τα από αυτές τις περιοχές αντί να απομακρυνθούν. Γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε καμία ε, οικονομία που να λειτουργεί στο Κογκό και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Είμαστε πολύ μακριά από τον Ντουτ Φρανκ. Ε, ξέρω ότι δεν ήταν τέλεια η νομοθεσία Ντουτ Φρανκ και πολλοί πιστεύουν ότι η Αμερικανική νομοθεσία οδήγησε σε ένα εμπάργκο de facto ε, είδαμε ύφεση της οικονομίας στο Κογκό, αλλά είδαμε ε, και πάλι να επανέρχονται εταιρείε και να κινείται η οικονομία. Τώρα το ότι υπάρχουν ε, στον Ανατολικό Κογκό κάποιες τέτοιες ε, πράσινες ε, περιοχές είναι επειδή υπάρχει ουσιαστικά υποχρεωτική νομοθεσία που ισχύει για όλους και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα πρέπει να αντιγράψει τι είναι σωστό και να μετακινηθεί μακριά από το τι είναι λάθος. Βέβαια, με καλούς σκοπούς δεν γίνονται τα πράγματα Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τα αριθμητικά στοιχεία που δεν ε, σέβονται τον Ντοντ Φρανκ. Ε, τελικά δεν κάνουν καμία προσπάθεια. Αν θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε στους Ευρωπαίους καταναλωτές ότι αγοράζουμε και πολλούμε προϊόντα που δεν προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές, θα πρέπει να στοχεύσουμε και στα καταναλωτικά αγαθά. Γιατί εδώ δεν εισάγουμε κυρίω πρωτεσίλε, αλλά καταναλωτικά αγαθά που παράγονται στην Νοτιοανατολική Ασία. Ε, τα iPad, τα κινητά, τηλέφωνα, όλα αυτά. Αυτά δεν παράγονται εδώ. Και αυτή τη στιγμή αυτά δεν καλύπτονται. Και νομίζω ότι θα ήταν και κάπως άδικο για τους ε, Ευρωπαίους αγωγείς πρώτων και τα ευρωπαϊκά χιτήρια να αφήσουμε άθικτη την μεγάλη καταναλωτική αγορά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ πολύ όλους που μας παρουσίασαν τις εισηγήσεις σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο συνέβη στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα. Απονείμαμε το βραβείο Ζαχάροφ σε έναν γιατρό από το Κονγκό που τον επεφημίσαμε και τον χειροκροτήσαμε όλοι όρθιοι επειδή κατέβαλε προσπάθειες ε, τους πιο ευάλωτους ανθρώπους να τους βοηθήσει σε αυτή την περιοχή. Συμφωνώ με την παρατήρηση, δεν είναι μόνο το Κονγκό, είναι όλες οι περιοχές σύραξης ε, παγκόσμια, αλλά όρθιοι τον χειροκροτήσαμε για αυτό, για τα αιτήματα που πρέπει να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα ακριβώς όπως αναφέρθηκε εδώ σε σχέση με την εξόριξη και εμπορία αυτών των μεταλλευμάτων και ορυκτών να είμαστε συνεπείς. Αυτή τη θέση να την εγγράψουμε νομοθετικά και να την κατοχυρώσουμε. Αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Και απηχώ και τις ε, παρατηρήσεις της Μαρίας για βιώματα και εμπειρία από άλλους τομείς. Για τον τομέα, για παράδειγμα, της μεταποίησης ε, προϊόντων. Πρέπει να μάθουμε και να συναγάγουμε τα ορθά συμπεράσματα. Και τέλος, ε, μια διασύνδεση όσον αφορά τη συζήτηση θεμάτων είπα. Διαρκώς μας λένε ότι TTIP δημιουργεί ένα νέο παγκοσμιοποιημένο οικουμενικό πλαίσιο και με μια νέα γεωδυναμική δυναμική. Αν συμβαίνει αυτό, αυτό θα είναι πραγματικά μια τεράστια συμβολική σημασία σε κίνηση όσον αφορά και τους πολίτες για το τι είναι η TTIP θα λέμε και θα τους πούμε ότι θέλουμε να αναβαθμιστεί η πολιτική εμπορίου μας ώστε να επιτευχθεί βελτίωση όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου και σε σχέση με το εμπόριο. Στη δική μας γεωγραφική επικράτεια, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, στη ΣΥΠΑ και παγκόσμια. Και αυτό είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο θα πρέπει να συνδέσουμε αυτά με τα οποία προαναφέρθηκαν. Να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα θετικά στοιχεία, επ' αυτό να οικοδομήσουμε με τη ΣΥΠΑ και να σημειωθεί πρόοδος επ' αυτόν και να υπάρχει μια δυνατότητα να είμαστε προπομπή εμείς πρωτοπόροι ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία λοιπόν που μας προσφέρεται. Να συνεργαστούμε ώστε να γίνει το επόμενο βήμα προς τα εμπρός και να μην οπισθοχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Η αίμα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους ε, τους αγορητές. Ε, εξαιρετικές ε, πληροφορίες μας έδωσαν όσον αφορά την εξόριξη αυτών των ορυκτών και μεταλλευμάτων. Πραγματικά βοηθούν για την εξέταση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα τύχει συνέχεια του χρόνου. Και ελπίζω ότι και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επίτροπη και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε με συμμετοχή των εμπλεκόμενων να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι θα κατανοήσουμε επιτόπου πώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι η πραγματικότητα όταν θα έρθει η ώρα και θα οριμάσουν και θα προχωρήσουν συζητήσεις για αυτό το θέμα. Υπάρχουν αρκετές παρατηρήσεις αλλά σε τρεις θα επικεντρωθώ. Κανείς δεν διαφωνεί ότι ουσιαστικά θα πρέπει να ολοκληρωθούν αυτές οι προσπάθειες. Συνεισφέρει η εξόριξη των ορυκτών στο να συνεχίσει η χρηματοδότηση για αυτές τις χώρες και οι περισσότερες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον σήμερα ότι σε σχέση με το εμπόριο των τριών τάφ και του χρυσού είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να μας κάνει να εξετάσουμε ποια είναι η καλύτερη οδός για να ενθαρρύνουμε να προχωρήσουμε προς την ορθή κατεύθυνση δεν είναι μόνο τα ορυκτά, το μόνο ζήτημα και ο μόνος ε, παράγοντας ε, για τα θέματα σειράξεων και την έκρηξη ε, βίας και έκρηθμη κατάσταση σε πολλές χώρες. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι θα εντάσσονται όλα αυτά σε μια ευρύτερη εικόνα και οι δράσεις μας. Αλλά φυσικά σε σχέση με την εθελούσια, εθελοντική δράση πρέπει να επικεντρωθούμε στην αλυσίδα τροφοδότησης. Και επειδή αναγνωρίζουμε σε σχέση με την τοποθέτηση ότι ακόμα και επιχειρήσεις που έχουν δεσμευτική προσέγγιση, ακόμα και στο μεταποιημένο προϊόν και με τις διατάξεις Don Frank δεν υπάρχει ουσιαστικά αυτή η απόλυτη ε, βεβαιότητα. Όλο και περισσότερες εταιρείες ε, λοιπόν όταν θέλουμε να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε και κάτι άλλο το οποίο δηλαδή αναγκάζουμε κάποιους ε, να ε, εγκαταλείψουν κάποιες χώρες επειδή υπάρχει κίνδυνος, κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν και έτσι αναγκάζονται να μετεγκατασταθούν και για τον ε, συνάδελφο που ανέφερε και με την δική του πείρα και είπε ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία τόπου αλλά και αρνητικά αναφέροντας αυτά και σε σχέση και με τις διακοιμάνσεις τιμών και για το Κονγκό και είπε ότι σταμάτησαν και εξορυκτικές δραστηριότητες. Αυτό είναι μια άλλη απειλή του να σταματήσουν, να τερματιστούν ε, οι δραστηριότητες αυτές. Όμως δεν θέλουμε να μείνουν άνεργοι οι άνθρωποι εκεί και να μείνουν ε, χωρίς απασχόληση. Πρέπει ε, να πούμε ότι δεν θα βοηθήσει καθόλου αυτό την κατάστασή τους. Πρέπει να βρούμε τους σωστότερους τρόπους για να δράσουμε. Και ακούσαμε επίσης ότι η υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ποσοστό λαθρεμπορίου. Και τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Να υπάρχει μια ισορροπημένη προσέγγιση. Να μην συνεισφέρουμε στο να εγκαταλείπουν κάποιες χώρες ε, εταιρείε ε, και οξυνθούν τα προβλήματα. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Με ποιο τρόπο μπορούν αυτές οι δράσεις και αυτές οι πρωτοβουλίες να ενταχθούν σε μια ενιαία εικόνα τι θα γίνει με την επιβάρυνση επιχειρήσεων. Θα υπάρξει έλεγχος για το, με, σχέση τη μία πρωτοβουλία με την άλλη νομοθετική δράση Don Frank. Πώς θα γίνουν οι έλεγχοι αυτοί ώστε να είναι λειτουργικοί και να μην παραμείνουν μη λειτουργικοί. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ε, ευχαριστία μου για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Δεν θέλω να καλύψω όλα τα σημεία, μόνο σε τρία θεματικά πλέγματα θα αναφερθώ. Μια και τίνω και εγώ επίσης υπέρ της ε, δεσμευτικής ρύθμισης, των δεσμευτικών ρυθμίσεων. Αλλά τίθεται μετά το ερώτημα αμέσως τι θα κάνουμε αν κάποιος δεν τηρήσει αυτά τα δεσμευτικά πλαίσια. Ποιες αντιδράσεις θα υπάρξουν, ποιοι μηχανισμοί προσφυγής ε, ή μηχανισμοί επιβολής μετακυρώσεων είναι ενδεδειγμένοι ώστε να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση. Διότι αν θέλουμε να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε αν κάποιος δεν συμμορφώνεται και δεν τηρεί αυτές τι διατάξεις. Θα ασκηθεί απλώς πίεση, πίεση θέση ή θα ασκηθούν και μέτρα ε, δικαίου, δηλαδή προσφυγή και ε, πρόστιμα ή κυρώσεις. Και για τα τέσσερα ορυκτά ουσιαστικά έχουν αυθαίρετα ε, επιλεγή επειδή προέρχονται από την περιοχή ε, και ε, αυτή των σειράξεων και στη μεταποίησή τους αντιμετωπίζουν αυτή την, αυτές τις Υπάρχουν όμως και άλλα τα οποία συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση ένοπλων σειράξεων. Χρειαζόμαστε σαφή κριτήρια. Αν δεν θέλουμε μακροπρόθεσμα να είναι αυθαίρετος ο χαρακτήρας και ο ρόλος με τον οποίο δρούμε και επιλέγουμε το ένα ή το άλλο και να μην βρίσκεται κάτω από ένα επίπεδο η εμπορική μας πολιτική όσον αφορά για παράδειγμα ε, κάποιο ε, κάποια επιβολή κυρώσεων. Έρχομαι στο τρίτο θεματικό σημείο, θεματολογικά. Πώς θα καθορίσουμε τις περιοχές σειράξεων ή με άλλα λόγια εκείνες τις περιοχές που θεωρούμε επίμαχες ζώνες. Επαρκεί το ανέφερε αυτό ένας αγορητής ε, σε σχέση με, τους, με τις επιχειρήσεις ε, να επιβάλλονται όροι και προϋποθέσεις ή θα πρέπει εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πούμε ότι θεωρούμε την μία ή άλλη περιοχή προβληματική και πώς μπορεί να ε, αναλυφθεί δράση επιτόπου ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Γιατί αυτό σε σχέση με μία ζώνη προβληματική σύραξης πρέπει να αποσαφινιστεί. Πρέπει να προβληματιστούμε περαιτέρω στην πρόταση της Επιτροπής και να βελτιώσουμε τα πράγματα για αυτού τους ορισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. θέλω και εγώ να κάνω μια-δύο ερωτήσει. Εγώ θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Αφενός ε, η σχέση Dodd Frank σε σχέση με μια ευρωπαϊκή ρύθμιση. Η αγορά ή το εμπόριο για παράδειγμα με αυτές τις πρώτες ύλες είναι θα λέγα περιορισμένη. Δεν είναι ατέλειωτες οι επιχειρήσεις που να δρούν σε αυτό το πλαίσιο. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν εξοικειωθεί όσες δρούν εκεί με τις διατάξεις Dodd-Frank και οι πελάτες επίσης ε, που ασχολούνται με την εμπορία αυτών των ορυκτών και ε, μια δεύτερη ρύθμιση από πλευράς ε, παράλληλης πλευράς δεν θα αποδυνάμωνε ίσως αυτούς τους μηχανισμούς και στην Global Witness στρέφομαι και διατυπώνω αυτή την ερώτηση. Όταν οικοδομούμε τόσο διαφορετικά συστήματα η μεν και η δε, το ένα μήπως αποδυναμώνει το άλλο. Και μια και σε σχέση εντωμεταξύ έχει ενταχθεί, έχουν ενταχθεί οι διατάξεις Dodd Frank ε, όσον αφορά τις σχέσεις με πελάτες και την εμπορία θα ήταν δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο και πώς θα μπορούσε να υπάρξει συμπληρωματική, παραπληρωματική δράση. Το δεύτερο το οποίο θέλω να ζητήσω, η άνηση μεταχείριση προϊόντων σε σχέση με την εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η το επισήμανε. Δεν μπορώ να το κατανοήσω ότι για παράδειγμα Κάποια προϊόντα είναι απόλυτα ελεύθερα από υποχρεώσεις και δεσμεύσεις ή περιορισμούς σε σχέση για παράδειγμα με άλλα πρώτες ύλες από ζώνες ε, ε, ένοπλης σύραξης. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια λύση του προβλήματος ε, μέσα σε ένα λογικό συγκρίσιμο πλαίσιο για τα μεν και τα δε. Και αυτό θα ήταν μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επίσης και προς τους πραγματογνώμονές μας. Α, ο κύριος Βίνκλερ, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, εσείς έχετε τον λόγο κύριε Βίνκλερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να προσθέσω και εγώ τη φωνή μου σε εκείνου που ευχαρίστησαν τους πραγματογνώμονες για όλες τις πληροφορίες που μας παρέσχαν σήμερα και για τις απόψεις που μας, ε, τις ιδέες που μας ε, έδωσαν. Είναι, ένα, είναι σημαντικό αυτό να έχουμε αυτές τις διαφορετικές κατευθύνσεις και προτάσεις ε, και σε σχέση με τα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου επικεντρωνόμενοι στο περιεχόμενο, στην ουσία της πρότασης. Είναι προφανές ότι πρέπει να βελτιωθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι επίσης πρόδειλο ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των διαφόρων εμπλεκομένων που παρίστανται σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Άλλοι επικεντρώθηκαν στο χαρακτήρα περισσότερο της ρύθμισης του κανονισμού λέγοντας ότι η εφαρμογή ή εθελοντικού πλαισίου, εθελούσιου πλαισίου ή υποχρεωτικού πλαισίου δεσμευτικού χαρακτήρα θα μπορούσε να επέλυε τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο χαρακτήρας δεσμευτικός ή όχι, αλλά το περιεχόμενο της ρύθμισης που πρέπει να δούμε αν θα επιλύει τα προβλήματά μας υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία με τα οποία πρέπει να ε, πορευθούμε. Συνάδελφος μίλησε για την ισορροπία. Πράγματι πρέπει να πετύχουμε μια προσεκτική ισορροπία μεταξύ των στόχων μας που είναι θεμητός ο στόχος για παράδειγμα του να διασφαλίσουμε την αηφόρο ανάπτυξη σε περιοχές υποσύραξη να διασφαλιστούν θέσεις απασχόλησης καθαρές ε, θέσεις ε, ε, εργασίας ε, και να μπορέσουμε στις σημερινές ζώνες σύραξης να δράσουμε, αλλά και τον άλλο πολύ σημαντικό στόχο που έχουμε και αυτό να τον λάβουμε υπόψη, που είναι να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας στην Ευρώπη, μέσα στο πλαίσιο ότι γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ στην στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του Συμβουλίου πρέπει να μεριμνήσουμε να διασφαλίσουμε αυτή την ε, συνεκτικότητα και συνοχή με τις θέσεις μας και τις δράσεις μας για την ανταγωνιστικότητά μας. Δύο θέματα από πλευράς μου θα χαιρόμουν αν θα μπορούσα να άκουγα από τον κύριο Ντίλαντ από τον ΩΣΑ για αυτές, αυτά τα στοιχεία που μας είπε για τον συμπληρωματικό χαρακτήρα, παραπληρωματικό ίσως χαρακτήρα μεταξύ όλων των πρωτοβουλειών αυτών. Και πώς γίνεται να επιτευχθεί αυτό, αν δεν είναι δυνατόν και αν είναι δυνατόν, ποια μέτρα θα μας συνιστούσε να εφαρμόσουμε. Και σημαντικό επίσης και η ελαστικότητα, η ευληγησία. Έχοντας παρακολουθήσει την ανάπτυξη αυτής της δυνατότητας με βάση την οδηγία αυτή, θα μπορούσε ίσως να μας επεξεργαστεί, να μας ε, αναλύσει περισσότερο πώς θα μπορούσαμε να δράσουμε ε, σε σχέση με τις προτάσεις του. Η άλλη ερώτηση φυσικά στρέφεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αδειμονώ να ακούσω πώς η Επιτροπή θα μπορούσε να εμπλέξει όλους τους εμπλεκόμενους και να υποβληθούν συγκεκριμένες εξειδικευμένες προτάσεις ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το στόχο μας με, επιτυχία. Ευχαριστώ. κυρία Μπεγκίνη Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια για την ομάδα EFTD Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές ε, και θα ήθελα και εγώ να βαθύνω σε κάποια θέματα στα οποία αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι Εβραίος. Καταρχήν, θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω το ότι ήδη έχουν υπάρξει εκούσια προγράμματα πιστοποίησης και μας ε, έχουν δείξει ότι ήταν αναποτελεσματικά καθώς οι φυσικοί πόροι συνεχίζουν να τροφοδοτούν ε, τις σειράξεις. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει σε ένα εκούσιο πρόγραμμα αν και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν επιλέξει ένα διαφορετικό καθεστώ και συμφωνώ με τον συνάδελφα που αναφέρθηκε στις ε, πιθανές ανισορροπίες ε, μεταξύ ε, ενός εκού συστήματος που κάποιοι θα μπορούσαν να υιοθετήσουν και κάποιοι άλλοι όχι και αναφέρουμε γιατί θα πρέπει μόνο να περιοριστούμε στα τέσσερα αυτά ορυκτά ενώ έχουμε και άλλα που τροφοδοτούν τους πολέμους. Κάτι ακόμη που θέλω να ρωτήσω. Γιατί περιοριζόμαστε σε κατέργαστα μεταλλεύματα και δεν μιλάμε και για μεταποιημένα μεταλλεύματα, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ε, ε, να χρησιμοποιηθούν και αυτά για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για τροφοδότηση σύγκρουσεων, αλλά θα θέλω κάποιες λεπτομέρειες ό,τι αφορά το ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην παραγωγική ελισίδα. Μπορείτε να μου πείτε ότι αν είναι υποχρεωτικό το σύστημα επιστοποίησης, ε, δεν ε, θα υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία και μεγάλο άχθος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Να μου πει ο εκπρόσωπος του ΕΣΑ πως ο ε, οδηγός δέωσης επιμέλειας θα σε λαμβάνουν υπόψη τη θέση μιας επιχείρησης στην παραγωγική αλυσίδα και αν πράγματι ένας υποχρεωτικός χαρακτήρας θα ήταν τόσο πολύ επιβαρυτική για τις μικρές και μεσέ επιχειρήσεις. Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα μπορεί να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο. Ναι, Πρόεδρε. Η κυρία Ράτσο βγήκε για ένα δευτερόλεπτο από, από την αίθουσα. Μπορούμε να προχωρήσουμε μετά τους ομιλητές. Καλώς. Τότε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράσεω, Χαούτιν. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να λάβω το λόγο για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Για την ε, παρουσίαση του κυρίου Μαλάση. Νομίζω ότι καθιστά σαφές ότι είναι πολύ περίπλοκη η πρόκληση η διάρρηξη του δεσμού μεταξύ των ε, περιοχών που πλήττονται από συγκρούσεις και της εξόρυξης των μεταλλευμάτων. Εδώ έχουμε να κάνουμε με επίλυση ε, διαφορών, έχουμε με χρηστή διαχείριση, με μεταρρυθμίσεις ως προς τις ροές αυτών των μεταλλευμάτων και της ε, αλυσίδας προμήθειας και διαφάνεια. Οποιαδήποτε τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να σημαίνει μια ευρύτερη λύση και για την περιοχή βέβαια των μεγάλων λιμνών, αλλά άλλωστε ο κανονισμός καλύπτει ένα ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο. Κάθε τέτοια λοιπόν ευρύτερη προσέγγιση σημαίνει προσχώρηση σε κάθε στοιχείο αυτής της προσέγγισης. Εμείς το κάνουμε αυτό. Μεμονωμένα, μία πρωτοβουλία διαφάνειας για την αλυσίδα προμηθειών από περιοχές που από συγκρούσεις δεν μπορεί μόνη της να λύσει μία σύγκρουση. Υπάρχει ο κίνδυνος πάντα της παραβίασης ή της διαφορετικής στάσης των επιχειρήσεων. Παραδείγματι, ακούσαμε στοιχεία για το ΙΣΚΙ, τον Κασίτερο και τη σχετική έρευνα από την Ρωμετό που μας λέει ότι είναι καθαρή η αλυσίδα. Αλλά δεν έχουμε καταγράψει, δεν έχουμε φτάσει μάλλον ακόμη στα προηγούμενα επίπεδα των εξαγωγών κασιτερίτη που ήταν για την τελευταία περίοδο στο ίμιση των εξαγωγών της περίοδου 2008-2009. Άρα είναι πολύ ευρύτερο το θέμα. Χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση. Και χαίρομαι για την, ε, για την παρατήρηση από Digital Europe ότι χρειάζεται μια σειρά από συνοδευτικά μέτρα. Ένα άλλο σχόλιο από κάποιον άλλον αμιλητή, ίσως βουλευτή αν θυμάμαι καλά, για την εκτίμηση του πόσα είναι τα μεταλλεύματα που εξορισόμενα μπορεί να συμβάλλουν στις ε, συγκρούσεις. Είναι ευρύτατος αυτός ο αριθμός. Γίνεται λόγος για ένα 13% από την ε, ε, από τον Οργανισμό Εθνών, αλλά για την ε, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, πέραν των μεταλλευμάτων, έχουμε και την ε, αλληλεία, έχουμε πολλές άλλες δραστηριότητες που φτάνουν μέχρι και τη φορολογία, πολλά μπορεί να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση μιας διαφοράς και ενόπλης σύγκρουσης. Πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν την αρχή της προσέγγισης με την αναγνώριση της πορείας ενός προϊόντος αλλά και της διαπεριφερειακής υποστήριξης του προγράμματος. Το ICGLR με την περιφερειακή ε, πρωτοβουλία για, τις, ε, για τους βιώσιμους πόρους και με ένα βιώσιμο μηχανισμό πιστοποίησης στην περιοχή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Για το θέμα των συγκρούσεων και των πληττωμένων περιοχών, τόσο εμείς όσο και η Επιτροπή, βλέπουμε ότι Θέλουν οι αρχές των κρατών μελών περισσότερες διευκρινήσεις ως προς το τι ορίζεται ως σύγκρουση. Αυτό ήδη το έχουμε τώρα στο άρθρο 2ε συμπεριλάβει του σχεδίου κανονισμού. Υπάρχει πολύ ευρέω δεδομένη γνώση, ανοιχτή και προσβάσιμη στο κοινό και από τη δική μας την υπηρεσία και από τα διάφορα think tank και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάνω απ' όλα να ζητούμε τους καλύτερους τρόπους αυτές οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες και στους φορείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτών. Να είναι διαθέσιμες για να μπορούν και μόνοι τους να αξιολογήσουν τον κίνδυνο και να μπορούν να τηρήσουν τις αρχές της δέουσης επιμέλειας για την προμήθεια, για την αλυσίδα προμηθειών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχήν, να πω δύο λόγια σε ό,τι αφορά γιατί επιλέγουμε την ακούσια προσέγγιση όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι αποτελεσματικό. Αναφέρθηκε αυτό το θέμα από πολλούς, από σου πήραν το λόγο. Κάτι που μάθαμε από τη δημόσια διαβούλευση και από τη μελέτη αντικτύπου και επίσης κάτι που αναφέρθηκε εδώ, από τον εκπρόσωπο της Digital Europe σήμερα ήταν ότι οι κατάντι εταιρείε ενδιαφέρονται στο να υπάρχει υπεύθυνη εξόρυξη μεταλλευμάτων γιατί δημιουργείται ισχυρή πίεση από τους καταναλωτές αλλά και από τον νόμο του Τράνκ. Παρ' αυτά, ξεκάθαρα έχουν συναντήσει δυσκολίες ε, επειδή είναι μακρές οι ελισίδες εφοδιασμού. Αν δούμε τώρα τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία τα λάβαμε από, την, από το πρώτο έτος της εφαρμογής της νομοθεσίας του Frank, μπορούμε να δούμε ότι μόνο 130 εκθέσεις ε, ε, ε, είχαμε, ενώ αναμέναμε 600 και πολλές εταιρείες δεν μπόρεσαν να καθορίσουν την προέλευση των μεταλλευμάτων στα προϊόντα τους και επομένως η διαφάνεια στο χιτήρια είναι θεμελιώδες και αυτός ήταν ένας από τους λόγους γιατί στην ευρωπαϊκή μας προσέγγιση ε, πήραμε διδάγματα από την ομοθεσία του Τφρανκ, από τη δέουσα επιμέλεια του ΟΣΑ. Επίσης, πήραμε διδάγματα και από τις θετικές και τις αρνητικές εμπειρίες. Επομένως, η πρότασή μας στο σχέδιο κανονισμού συμπληρώνει το νόμο του Τφρανκ. Βασίζεται τα μάλα στη ε, δέουσα επιμέλεια του ΟΣΑ ουσιαστικά δεν είναι ο σαμίων, αλλά ο σασίν. Καταρχήν δημιουργεί ένα κατάλογο χιτηρίων και εδώ θα ήθελα να απαντήσω σε όσους ρώτησαν τι γίνεται με την ανταγωνιστικότητα και αν θα στοχεύουμε μόνο τα ευρωπαϊκά χιτήρια. Όχι, δεν θα στοχεύουμε μόνο στα ευρωπαϊκά χιτήρια, αλλά παγκόσμια χιτήρια. Έχουμε ευρωπαϊκό κατάλογο, αλλά θα περιλαμβάνει τα χιτήρια παγκοσμίω που σέβονται τις δικές μας απαιτήσει. Και ε, σέβονται και τη δέουσα επιμέλεια πιστοποίησης. Τώρα, αυτός ο λευκός κατάλογος ε, θα κατονομάζει όσους λείπουν, αλλά θα ε, υπάρχει και πλήρης διαφάνεια στην αλυσίδια εφοδιασμού και φυσικά αυτό θα ωφελεί και τη διαδικασία της επιχειρήσεις κατάντι. Οι επιχειρήσεις κατάντι μπορούν να, να βασιστούν επίσης το σύστημα πιστοποίησης των εισαγωγέων και μπορούν και να βασιστούν σε αυτόν τον κατάλογο, τον λευκό κατάλογο των χιτηρίων. Σε σχέση τώρα ε, με την ερώτηση του Σιγητή Γουίνκλερ πώς μπορεί να συνεργαστεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μερικομισιών για να φτάσει πιο κοντά στο στόχο το σχέδιο κανονισμού δεν ε, είναι ένα έγγραφο που στέκεται από μόνο του, Συμπληρώνονται από συνοδευτικά μέτρα τα οποία υπάρχουν στην ανακοίνωση, το χάρη δημόσιες συμβάσεις που ε, θα ε, στοχεύουν στις καταντεπιχειρήσεις όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσμίω δηλαδή όσους θέλουν να συμμετέχουν, ω εισαγωγή θέλουν να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς. είναι κίνητρα λοιπόν. Επίση, υπάρχει τεχνική και οικονομική βοήθεια στι μικρέ και επιχειρήσει. επιχειρήσεις. Ε, άκουσα πολλού που υπογράμμισαν τη σημασία αυτών. Και επίση ε, θα υπάρχει και μια χρηματοδότηση στα χιτήρια ε, για να υθετήσουν το πρόγραμμα και θα υπάρχει και πολιτικός διάλογος. Επομένως βλέπετε ότι τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν στη διαδικασία. Τώρα, εδώ θα ήθελα να αναφερθώ και στις νέες εξελίξεις από τότε που παρουσιάστηκε η νέα πρόταση, η αποκάλυψη των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Αυτό είναι κάτι που ήδη υφίσταται και στοχεύει τις εταιρείες ε, και τις ενθαρρύνει να υποβάλουν εκθέσεις. Πρέπει να δούμε βέβαια και το πλαίσιο. Υπάρχουν ε, και άλλα μέσα και άλλα νομοθήματα που ε, αναφέρουν ε, αυτή την ε, δημοσιοποίηση. Έχουμε τη διαφάνεια στις πληρωμές των εξορρυκτικών βιομηχανιών. Όλα αυτά θα είναι αλληλοσυμπληρούμενα. Για το θέμα του ελέγχου, auditing, η πρόθεση είναι να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα λογιστικού ελέγχου που θα βασίζεται στα πρότυπα του ΩΣΑ οι ελεγκτές και οι εισαγωγείς θα μπορούν να βασίζονται σε αυτό και θα πρέπει ε, να λαμβάνονται υπόψη τα ίδια υφιστάμενα προγράμματα για τις βιομηχανίες. Και κάτι τελευταίο, αλλά επίσης σημαντικό, γιατί δεν έχουμε αντιγράψει τον Αμερικανικό νόμο Dodd Frank. Κάποιοι ομιλητές αναφέρθηκαν στην ε, ανάλυση του αποτελέσματος του σοκ που δημιουργείται και ότι υπάρχει και διαφοροποίηση του εμπορίου. Απουσία επαρκούς ε, ικανότητας για υπεύθυνη εξόριξη μεταλλευμάτων στις εμπόλεμες ζώνες και επίση, ε, έχοντας κατά νου ότι ο δικός μας κανονισμός έχει ένα παγκόσμιο πεδίο, δεν καλύπτει μόνο την περιοχή των μεγάλων λιμνών όπως η νομοθεσία του Φρανκ. Η προσέγγιση μας ε, συνάδει με τον ΩΣΑ. Επομένως, αν δεν υπάρχει επαρκή ικανότητα που είναι εύκολο για τις εταιρείε να φύγουν και να βρουν άλλες συναλλακτικές. και στην ε, έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμένων του ΙΕ διφάνει ότι στο Κογκό υπάρχει λαθρεμπόριο ε, ορυκτών, κυρίως του χρυσού και αυτό έχει αυξηθεί και φυσικά χάνονται θέσεις εργασίας και φορολογικά έσοδα και φυσικά αυτά δεν είναι τα αποτελέσματα που θα θέλαμε να έχουμε. Νομίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις που τέθηκαν από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Έχω και μια ερώτηση περαιτέρω για το πώς θα χρησιμοποιηθούν οι δημόσιες συμβάσεις ως κίνητρο για τις εταιρείε για να διαθετήσουν το οικοσύστημα. Αλλά κατόπιν θα πρέπει να αλλάξετε τον κανονισμό για τις δημόσιες συμβάσεις, έτσι δεν είναι. Όχι, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Για τη νέα οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες που 2024 εε επιτρέπει, ναι, επιτρέπει απλώς όμως, δεν το καθιστά επιτακτική ανάγκη, δεσμευτική υποχρέωση, Α, μάλιστα, όχι λέει ο ομιλήτρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΕ και σίγουρα το Ευρωκοινοβούλιο είναι κάτι που δεν ενθάρρυνε σε σχέση με το να υιοθετηθεί αυτό το υπόδειγμα. Είναι κάτι που τα κράτη-μέλη μπορούν αν επιθυμούν να συμπεριλάβουν και θα ενθαρρύναμε να συμπεριλάβουν στις ρήτρε αυτές για τις δημόσιες προμήθειες αυτό το χαρακτήρα. Εντάξει, ωραία, πολύ καλά. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στους ε, πραγματογνώμονες. Την δυνατότητα σύντομα να απαντήσουν περιεκτικά και πρώτα απ' όλα ο εκπρόσωπος του ΩΣΑ παρακαλώ. έχει τον λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τα πολύ θετικά σχόλια και τις παρεμβάσεις που ακούσαμε, σήμερα. Είναι σαφές ότι το Κοινοβούλιο ε, με μεγάλη κέρια σημασία που δίνει σε αυτά τα θέματα και το ρόλο του, προτού επισέλθω στο συγκεκριμένο ερώτημα, θεωρούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κοινή ανακοίνωση για αυτά τα μέτρα. Θεωρούμε ότι πράγματι θα βοηθήσει να υπάρξουν κίνητρα για την ε, πρωτοβουλία του ΩΣΑ για την, τον αποτελεσματικό χαρακτήρα και να αποφύγουμε αρνητικές επιπτώσεις ή εμπάργο. Είναι λοιπόν χρήσιμη αυτή η πρωτοβουλία για τις δημόσιες προμήθειες και έχει κέρια σημασία για την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών. Θεωρούμε ότι τα συμπληρωματικά μέτρα από κοινού θα έπρεπε βήμα προς βήμα κλιμακούμενα να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται με το σχέδιο κανονισμού. Υποστηρίζουμε αυτή την προσέγγιση. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της πρότασης, φυσικά θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο κύριοι ε, στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν. Πρώτα απ' όλα η αποτελεσματικότητα σε σχέση με τον ε, ε, δεσμό διασύνδεση περιοχής σύραξης και αυτών των ορυκτών. Το δεύτερο, να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείε στην Ευρώπη που θα χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα θα είναι υπεύθυνε και αυτό είναι ένας στόχος. Αναφέρθηκε και έχουν θεσπιστεί αρχές για την υπεύθυνη εταιρική δράση. Είναι ένας στόχος λοιπόν αυτός αφ' αυτού ότι οι εταιρείε αυτές θα έπρεπε να δρουν με υπεύθυνο τρόπο, με εταιρική υπευθυνότητα. Δεν είμαστε εμεί σε θέση να συστήσουμε πιο συγκεκριμένα αν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα ή εθελοντικού χαρακτήρα. Ξέρουμε ότι η σύσταση αυτή σε σχέση με την υιοθέτησή της και την πολιτική βούληση που συνεπάγεται για να υιοθετηθεί. Φυσικά υπάρχουν δυνάμεις της αγοράς υπό το 1502 τμήμα του, του νομοθετήματος Dodd Frank που θα ε, ήθελαν να υπάρξει το πλαίσιο opt-in σε ένα εθελοντικό πλαίσιο. Όμως η, η δεσμευτική ρύθμιση θα απέστελε ένα πιο ισχυρό μήνυμα ε, συνολικά. Εμείς πιστεύουμε ότι εφόσον αυτή η πρόταση και η πιστοποίηση θα σχεδιάζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ και θα υπάρχει εθελοντικός χαρακτήρας και θα διασφαλίζεται ιδέωσα αμέριμνα που πρέπει να ε, διασφαλίζεται, ε, τότε αν συνδεθούν αυτά τα συμπληρωματικά μέτρα με αυτά τα στοιχεία θα είμαστε αποτελεσματικοί. Για την ερώτηση συγκεκριμένα για την ε, συμπληρωματικότητα με το νομοθέτημα, με το νόμο Dodd Frank. Ε, και σε σχέση με επικαλύψεις ρωτήθηκε. Η απάντηση όχι. Αλλά εξαρτάται ποιοι θα είναι ακριβώς αυτοί οι κανόνες και ρυθμίσεις. Ε, αν θα βασίζονται στις κατευθυντήρες γραμμές ως πρότυπο του ΩΣΑ, όπως ε, σε κάποιο βαθμό η Dodd Frank επιβάλλει στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούνται τα πρότυπα του ΩΣΑ όταν υποβάλλονται εκθέσεις και ε, υποβάλλονται τα στοιχεία τους και οι περιφερειακοί μηχανισμοί διαπίστευσης και πιστοποίησης βασίζονται σε αυτές τις ε, κατευθυντήριες γραμμές του ΩΣΑ και έτσι λειτουργούν. Υπάρχει λοιπόν ένα κοινό πεδίο δράσης, ε, ένας κοινός παρονομαστής εκεί και γι' αυτό εμείς θα θέλαμε αυτές οι οδηγίες κατευθυντήριες γραμμές του ΩΣΑ να ακολουθούνται. Αυτό θα σημαίνει όμως ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στα χιτήρια. Αν αρχίσουμε και αναμένουμε περισσότερες, ε, περισσότερους ελέγχους ε, σε διαφορετικά περισσότερα επίπεδα αυτό θα δημιουργήσει σύγχυση και θα είναι αναποτελεσματικό. Θα πρέπει σε όλη την αλυσίδα λοιπόν τροφοδότησης να λαμβάνετε αυτό υπόψη. Τώρα σε σχέση με τα προγράμματα τα οποία θα είναι σημαντικό να ενταχθούν και να μπορέσουν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους. Η επιτήρηση λοιπόν, η εποπτεία και η συμμόρφωση, η επιβολή των κανόνων και κανονισμού πρέπει να διασφαλίζεται με έναν τρόπο συνεπή και συνεκτικό με τις ε, οδηγίες του ΟΣΕ. Σήμερα από πλευρά ΩΣΑ δεν υπάρχει κάποια προσπάθεια εποπτείας αυτών των μηχανισμών και δραστηριοτήτων, αλλά ίσως μπορεί να επιτελεστεί στο μέλλον αυτό. Τώρα για τις εκθέσεις και ε, την κατάθεση αναλύσεων ε, οι οδηγίες λένε με σαφήνεια πώς μπορούν για την δέουσα μέρημνα και επιμέλεια οι εταιρείε να υποβάλουν τα πορίσματά τους και τα στοιχεία τους. Θα είναι διαβαθμισμένες πληροφορίες αυτές εμπιστευτικού χαρακτήρα ε, μέσα στο πλαίσιο της τροφοδοσίας. Αναμένουμε να υποβάλουν στοιχεία για τις διεργασίες και διαδικασίες οι εταιρείε. όχι αναγκαστικά εξειδικευμένα ε, ε αναλυτικά στοιχεία θα ήθελα ένα πράγμα να υπογραμμίσω που έχει μεγάλη σπουδαιότητα για να κατανοήσουμε το θέμα της ε, δέουσας ε, επιμέλειας. Είναι ιδιαίτερη ευθύνη και πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες από τις επιχειρήσεις για να καλύπτεται αυτό. Αν είναι λοιπόν ε, υλικό από μια ε, ε, περιοχή σύρεξης θα πρέπει να υποβάλλονται τα στοιχεία αυτά. Αν όμως προέρχεται από μια χωρίς σειράξεις ε, ε, περιοχή, όμως θα μπορούσε να συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο λόγω για παράδειγμα εγκληματικών δραστηριοτήτων εκεί. Γι' αυτό επειδή δεν θέλουμε να ενθαρρύνουμε μια κατάσταση όπου θα καλύπτουν οι εταιρείε ε, την υποχρέωσή τους αυτή μόλις θα βρίσκονται σε ένα σαφές ε, ε, προσδιορισμένο πεδίο δραστηριοτήτων και μετά όταν θα εξέρχονται αυτού δεν θα επομίζονται πλέον, δεν θα επιβάλλεται σε αυτές τέτοιος περιορισμός. Θα θέλαμε λοιπόν μέσα σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο να υποβάλλεται αυτή η πληροφόρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο κύριος Μαλάση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα την κυρία Αρένα η οποία κάλεσε τους βουλευτές να κάνουν τον παραλληλισμό με την πορεία των γεωργικών προϊόντων χρησιμοποιώντας τρόφιμα. Είναι ακριβώς παράλληλες οι πορείες. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι οποιοδήποτε μέτρο θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να παρακολουθεί το τι εφαρμόζεται, γιατί πάντα κάποιος υπάρχει που θα προσπαθήσει να ε, ξεφύγει από, ε, από τον έλεγχο, είτε είναι θελοντική η συμμετοχή. Ε, έχουμε παραδείγματι υπηρεσίες ή επιχειρήσεις πιστοποίησης προϊόντων που εξορίσονται από την κόκκινη λεγόμενη ζώνη στο Κούγκου, ή στην Ουρίλ ε, και δίνουν πιστοποιητικό από πράσινες ζώνες. Αυτές οι επιχειρήσεις μοιράζονται τα έσοδα με τις πολιτοφυλακές. Στέλνουν τα χρήματα στη Σαμπούντα, δηλαδή στο δημόσιο ταμείο, νομιμοποιώντας έτσι αυτό το παράνομο χρήμα. Και έτσι παραποιώντας ακόμα και συμπληρωματικά μέτρα, γιατί αυτά χρειάζονται να υπάρχουν, ε, η παρακολούθηση από τη δικαιοσύνη και η επαλήθευση ότι τα γεγονότα που δηλώνονται όντως έχουν λάβει χώρα. Ε, θα ήθελα να πω επίσης ότι η νομοθεσία Dodd Frank δεν έχει φέρει αρνητικά αρνητικές συνέπειες. Μπορεί να δόθηκε και αυτή η εντύπωση στην αρχή, αλλά χάρη σε αυτή την πίεση τώρα μπορούμε να κάτσουμε ε, στο ίδιο τραπέζι με τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων και να συνομιλούμε. Χάρη σε αυτή την νομοθεσία σε κάθε επαρχία θεσπίστηκαν οι επιτροπές ελέγχου. Χάρη σε αυτή την νομοθεσία γίνεται η προσπάθεια της πιστοποίησης των ορυχείων, της διαδικασία πιστοποίησης των προϊόντων και Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να επιταχυνθούν και σε παγκόσμια κλίμακα. Έτσι μπορείτε να στηρίξετε άλλωστε και την, ε, τις ενισχύσεις που προσφέρετε σε άλλους τομείς. Όπως σε παραδείγματι στις εκλογές. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι οι εκλογές θα φέρουν κάποια άλλαγη ή ότι θα έχουμε καλή χρηστή διοίκηση εάν συνεχίζονται αυτοί οι πόλεμοι ή εκτοπισμοί του πληθυσμού. Το 5% μου λέτε είναι λίγο, μα και μία ανθρώπινη ζωή να σωθεί θα αρκούσε. Αν μπορέσετε λοιπόν να επιβάλλετε αυτήν την νομοθεσία και αυτή ε, και από την πλευρά της και η νομοθεσία Dot Frank αν μπορούσε να φέρνει αποτελέσματα, να τεθεί σε λειτουργία τουλάχιστον η διαδικασία. Πρέπει να τολμήσουμε, πρέπει να προσπαθήσουμε και ε, σας διαβεβαιώ ότι η κοινωνία των πολιτών θα σας είναι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κύρον. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα συνεχίσω σε αυτά που είπε ο κύριος Μαλαζή η συνειδητοποίηση έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά και τα αποτελέσματα επιτόπου που έχουν τεράστια ε, θεμελιώδη σημασία, γιατί αφορούν όχι μόνο την αλυσίδα της ε, πρόσθεσης αξίας, ε, δηλαδή την εξόριξη, το χιτήριο, τον εξευγενισμό, την παραγωγή και κατεργασία του προτελικού προϊόντος, αλλά όλου του τοπικού φορεί του οποίου εμεί δεν μπορούμε να επηρεάζουμε. Άρα χρειάζονται και τα συνοδευτικά μέτρα για να προβληθεί ο δικό του ρόλος και να δοθούν οι σχετικέ απαντήσει. Τώρα ε, στιγματίζονται τα ε, μεταλλεύματα με τα τρία τι και χρυσό που καταδικάζονται γιατί μιλάμε όμω για την περιοχή του Κονγκό γιατί αν μιλούσαμε για άλλε περιοχέ πληττόμενε από συγκρούσει και για άλλα μεταλλεύματα θα μιλούσαμε αλλά και για άλλα τελικά προϊόντα. Άρα χρειάζεται να κάνουμε τις σχετικές τις συνδέσεις. Για της κυρία Αργεντίνη, που ίσως επισημαίνει κάτι που δεν αντελήφθη από την έκθεσή μου για την έλλειψη κινήτρων για τα χιτήρια. Δεν εννοούσα εγώ αυτό. Εγώ εννοούσα ότι δεν υπάρχουν κίνητρα για τη φάση μετά τα χιτήρια, γιατί καλύπτονται τα χιτήρια είτε με την Dot Frank είτε με τα εθελοντικά προγράμματα καλύπτονται. Συμφωνώ απολύτως με την κυρία Σαρτζεντίνη ότι πρέπει να ακολουθήσουμε ε, τα μέτρα που φέρουν αποτελέσματα και να αφήσουμε αυτά που δεν φέρνουν. Σε θελοντικό επίπεδο, σε επίπεδο ε, αποτελεσμάτων των προγραμμάτων του ΩΣΑ, όπου βλέπουμε να έχουν καλά αποτελέσματα, ας τα παρακολουθήσουμε, ας τους δώσουμε συνέχεια, ας εντοπίσουμε την πεμπτουσία τους, τη θετική τους πεμπτουσία, ας συμπληρώσουμε με συμπληρωματικά μέτρα και συνοδευτικά μέτρα της Επιτροπής και έτσι ας εξασφαλίσουμε ότι δεν θα προκύπτουν αντίξωα ή ανεπιθύμητα αποτελέσματα και κυρίως όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Ε, επίσης για να επανέλθω στην κυρία Αρενά, βεβαίως και είναι επίκεντρο ουσιοδέστατο επίκεντρο όλων των επιλογών και ε, διαβημάτων του κλάδου η ανθρώπινη ζωή. Επειδή γνωρίζαμε τα προβλήματα, κάναμε τις προσπαθίες μας, μας για να δώσουμε απαντήσεις. Ως προς τα μέσα που έχουμε στη θέση μας τώρα, κάποιες επιτυχίες εξασφαλίζονται και χάρη στα προγράμματά μας αποδεδειγμένα, άλλωστε και με στατιστικές των τοπικών αρχών και πάλι με την επισήμανση σε παρένθεση του φαινομένου της ευθοράς μπορεί να συνδέεται με αυτό, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και αριθμητικά στοιχεία που μπορούν να αποδείξουν αυτή την ε, επιτυχία. Εάν θέλετε πιο πολλά στοιχεία, έχουμε από τον τομέα των κρατικών υπηρεσιών μια συνάδελφο εδώ που μπορεί να σας δώσει πιο πολλές λεπτομέρειες. Η ανταγωνιστικότητα όμως είναι κέρια σημασίας γιατί η επιτυχία αυτών των επιχειρήσεων εδώ στην Ευρώπη και των Ηνωμένων Πολιτειών βεβαίων αντίστοιχα των επιχειρήσεων ε, είναι δυνατή επειδή βρίσκονται οι επιχείρησεις αυτές στην αγορά και επειδή παραμένουν ανταγωνιστικές. Εάν όμως τις υποχρεώσουμε σε μια πορεία που δεν θα τους επιτρέπει τη διαφύλαξη της, ανταγωνιστικότητά της ανταγωνιστικότητάς τους, τότε ακριβώς κινδυνεύουμε να χάσουμε την πορεία αυτή και την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Για το εθελοντικό σύστημα πολλά υπόθηκαν. Νομίζω ότι το εφιστάμενο αυτή τη στιγμή εθελοντικό σύστημα με τα μέτρα που συνοδεύουν είναι de facto υποχρεωτικό γιατί όπως ανέφερε και ο συνάδελφος οι επιλογές της αγοράς υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χιτηρίων, σε επίπεδο μονάδων εξευγενισμού να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές. Άρα το ζήτημα που πρέπει να κρυθεί δεν είναι αν θα είναι θελοντικό ή υποχρεωτικό το σύστημα. Είναι να υπάρχει η επιτόπου στις περιοχές αυτές παρακολούθηση, η ε, συμπλήρωση με τα συνοδευτικά μέτρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Λακάρτ. Να ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουν τοποθετηθεί ε, υπέρ ε, της αποτελεσματικότητας ε, του νόμου Dodd Frank και επίσης ε, θα δούμε και τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας για το Τουγκστένιο και τα Λεμέτελα. Αυτά είναι πλήρη προγράμματα που έγινε πάρα πολλή δουλειά για αυτά και θέλω να ευχαριστήσω και τον τομέα των μεταλλευμάτων καθώς υιοθέτησε τη δέουσα επιμέλεια, έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες και νομίζω ότι συλλογικά αρχίζουμε να βλέπουμε να γεννώνται αποτελέσματα από τις προσπάθειες. Προφανώς ε, υπάρχουν αυτές οι πρωτοβουλίες και γι' αυτό είπα ότι είναι απολύτως σημαντικό να έχουμε μια επιπρόσθετη τεχνική συζήτηση για να δούμε λεπτομερώς τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν και να σχεδιάσουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα που να συμπληρώνει αυτά που ήδη υπάρχουν και να μην ε, τα αντιφάσκει. Και φυσικά θα πρέπει να δούμε και τον ε, οικονομικό αντίκτυπο της νομοθεσίας ε, Dodd Frank έχει βελτιωθεί η οικονομική δραστηριότητα και φυσικά έχει σχεδιαστεί για να ε, βοηθήσει τους ανθρακορύχων που ζουν ε, στα ορυχεία με τις οικογένειές τους. Ε, περί αυτού πρόκειται, πρόκειται για το να έχουμε υπεύθυνη δράση, αλλά συνεχίσουμε και να δραστηριοποιήμαστε στην περιοχή. Εγώ νομίζω ότι τώρα προστίθεται την Ευρωπαϊκή Ένωση αξία σε αυτό με την πρωτοβουλία συγγνώμη, με τις πρωτοβουλίες και την νομοθεσία Dot Frank έχει σταλεί ένα τεράστιο μήνυμα στην αγορά και φυσικά σε εταιρείε όπως η δική μου έχουμε και ενδιαφερόμενα μερέλη και μετόχους που συνεχώ πιέζουν τις εταιρείε να εξετάζουν την αλυσίδια εφοδιασμού και να εξαλείψουν ε, ε μετάλλα από τέτοια προέλευση. Έτσι λοιπόν, Φυσικά και προστίθεται αξία από την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, γιατί η νομοθεσία του Φρανκ ενώ επικεντρώνεται στο Κογκό και στις γύρω περιοχές, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία έχει ευρύ γεωγραφικό πεδίο. Και πάλι όμως, ε, τι εννοούμε με αυτές τις ζώνες υψηλού κινδύνου, με ε, Πρέπει να το ορίσουμε πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί να ορίσουμε μία ζώνη σειράξεων, αφού γίνει ορισμός, μόνο τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε τα συστήματα να, και μόνο τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε συστήματα ενχνασιμότητας ε, για ένα χιτήριο, το χάρη, χρειάζεται περίπου ένας χρόνος. Πρέπει λοιπόν ε, να είμαστε ευέλικτοι, ε, μιλήσαμε και για ανάντι και κατάντι εταιρείε. Εμείς ε, επίσης αναφέραμε τις δυσκολίες πόσο δύσκολο είναι να φτάσει κανείς στην αλυσίδα εφοδιασμού γιατί έχουμε χιλιάδες εφοδιαστές. Έτσι λοιπόν γι' αυτό μιλάμε για το επίπεδο των χειτερίων. Υπάρχει μεγάλη πίεση στις εταιρείες. Είναι ευθύνη των εταιρείων να στείλουν σημάδια πάνω και κάτω στην αλυσίδα εφοδιασμού. Όμως πρέπει να τους δώσετε ευελιξία και πρέπει να δώσετε ευελιξία σε εταιρείε για να κοινοποιήσουν πώς επικοινωνούν καλύτερα με τους προμηθευτές αλλά και με τους πελάτες τους. Νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ για το υποχρεωτικό τώρα ή εκούσιο χαρακτήρα νομίζω ότι είναι κάπως νωρίς να καταλήξουμε σε συμπέρασμα. Έτσι λοιπόν περιμένουμε να γίνει μια συζήτηση τεχνικού χαρακτήρα πρώτα. Ευχαριστώ. Και τέλος ο κύριος Γκίπ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σύντομα να ανταποκριθώ σε κάποιες από τις παρατηρήσεις που έγιναν. Πρώτα να αναφέρω ότι ακούσαμε πολλά, γιατί πολλές ε, από τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες ε, των επιχειρήσεων σε σχέση με τις δράσεις της ΕΠΑ και σε σχέση με την, ε, το νομοθέτημα Lord Frank θα θέλαμε να δοθεί ιδιαίτερη προώθηση σε σχέση με προτάσεις ε, για τις επιχειρήσεις αυτές ε, όσον αφορά την αντιμετώπιση των υλικών, των πρώτων υλών από περιοχές κινδύνου. Ακούσαμε και για τους καταναλωτές και η ανάγκη καταναλωτών να υπάρχουν εγγυήσεις ότι τα προϊόντα τα οποία θα αγοράζουν δεν θα τους εμπλέκουν σε τέτοιου είδου σειράξει. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναφερθεί το ότι δεν είναι η ευθύνη των ε, ε, καταναλωτών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει στις επιχειρήσεις κάτι τέτοιο. Παραμένει ευθύνη των επιχειρήσεων να διασφαλίζουν αυτή την πτυχή έναντι των καταναλωτών. Ακούσαμε επίσης για νέους κινδύνους αγορών και θα ήθελα εδώ να αναφέρω αυτό το οποίο ανέφερε πιο πριν η ΟΣΑ ότι αυτό δεν είναι για μια εγγύηση 100% ότι όλα θα είναι απόλυτα στεγανά και τέλεια. Είναι διαδικασίες που θα διευκολύνουν να διασφαλίσουν οι εταιρείε ότι κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους ώστε οι κίνδυνοι αυτοί να ελαχιστοποιούνται. Και σίγουρα αυτοί δεν είναι νέοι καινούργοι κίνδυνοι. Είναι ε, κίνδυνοι που αφορούν την τροφοδότηση των, ε, ε, της αλυσίδας τροφοδότησης και πολλές φορές υπάρχει έλλειψη υπαρκού ζήλου και επιμέλειας ώστε να διασφαλίζεται αυτή η ανάγκη είναι και το θέμα για παράδειγμα και άλλων υλικών που μπορεί να χρηματοδοτούν τέτοιου είδους σειράξεις και υπάρχουν ε, και ε, φήμες ε, για τέτοιου είδους υλικά παράλληλα με τα τρία τάφ και τον χρυσό που μπορεί τέτοιου είδους όπως τα σμαράγδια για παράδειγμα στο Αφγανιστάν και άλλα, άλλοι πολύτιμοι λίθοι που προέρχονται από την Κολομβία, χώρες της Αφρικής. Υπάρχουν λοιπόν και άλλες πολλές χώρες και περιοχές όπου θα πρέπει να ασκείται δέουσα επιμέλεια με τον τρόπο που απαιτούμε. Και η προσδοκία που υπάρχει ότι οι εταιρείε θα είναι προσεκτικές και θα ασκούν στο μέγιστο βαθμό την ε, επιμέλεια με ζήλο από πλευρά τους ε, για να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι. Και θα ήθελα επίσης να προσθέσω ε, δύο λόγια για τις τοπικές επιπτώσεις του νόμου Ντόρ Φρανκ. Έχει σπουδαιότητα να αναγνωρίσουμε και γι' αυτό το ανέφερα εισαγωγικά αυτό, το ότι ε, η κατάσταση δεν μπορεί να διατηρηθεί πλέον ε, περαιτέρω. Πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει μεγαλύτερη διεύρυνση αυτών των προβλημάτων και των σειράξεων. Και να ε, ε, αντιμετωπιστεί όπως πρέπει η ανάγκη επιμέλειας. Ε, είναι ιδιαίτερα περίπλοκες οι τριβές αυτή τη στιγμή και πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι δυνατόν με απλουστευτικές λύσεις να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Αυτά που είδαμε είναι μια σύνθετη εικόνα με έναν αριθμό θετικών αποτελεσμάτων. Πρέπει να αυξηθεί η επιτήρηση και η παρακολούθηση Όσο αφορά την εξόριξη αυτών των ε, αγαθών. Δεν υπάρχει μια σαφής εικόνα για όλα αυτά τα προϊόντα. Ακούσαμε ότι ε, για παράδειγμα για κάποιες περιοχές ε, και επαρχίες που υπάρχουν προβλήματα και σε σχέση με την ε, ε, το εμπάργο για το, για Κονγκό που ε, το, διαφοροποιείται η κατάσταση από επαρχία σε επαρχία και από περιοχή σε περιοχή. Ακούσαμε στην απαγόρευση, προεδρική απαγόρευση εξόριξης προϊόντων, π.χ. για το Κίβου, καθώς επίσης και για τις δραστηριότητες που λαμβάνονται για να διαφοροποιηθούν οι διαδικασίες σχέση με τις διαδικασίες Dodd-Frank. Και για να απαντήσω τελικά αν σε σχέση με την πρόταση του ΩΣΑ θα αποδυναμωνόταν το ο νόμος Dodd-Frank. Εφόσον υπάρχει ευθυγράμμιση με τις ε, διατάξεις ε, του ΟΣΑ, οι άλλες πρωτοβουλίες μπορεί να είναι συμπληρωματικές μέσα στο πλαίσιο του Dodd-Frank και να διασφαλίσουμε ότι θα καλύπτονται περισσότερες επιχειρήσεις από ό,τι σήμερα και έτσι να δημιουργηθεί μια προώθηση της ε, ενίσχυση της αρχής ε, ε, της ε, δέουσας επιμέλειας και να αυξήσουμε έτσι τη μόχλευση που έχουμε τη δυνατότητα άσκησης επιρροής στις, στις δραστηριότητες των χιτηρίων και στην τήξη των μετάλλων αυτών θεωρούμε ότι είναι η ευθύνη όλων των επιχειρήσεων ε, να μπορούν να επιβάλλουν την αρχή και να σέβονται την αρχή της δέουσας επιμάλειας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ε, επαΐοντες ε, που συνεισέφεραν με τις προτάσεις τους προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα ο κύριος Βίνκλερ θα λάβει τον λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ αγαπητοί φιλοξενούμενοι και αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω κάναμε ένα βήμα προς τα εμπρός σήμερα. Αποσαφηνίσαμε κάποια πράγματα. Όπως επίσης πιστεύω ότι αποσαφηνίσαμε ότι υπάρχει μακρύς κατάλογος θεμάτων που πρέπει ακόμα περαιτέρω να συζητηθούν μεταξύ μας. Και νομίζω ότι όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα έχουν συνειδητοποιήσει ότι η διάρκεια και τα συνοδευτικά μέτρα είναι πολύ μεγάλη σπουδαιότητα Αν σε σχέση με πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε στο να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, οι προσπάθειές μας πρέπει να συνεχιστούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει το δυναμικό αυτό να αναπτυχθεί από πλευράς των εμπλεκόμενων και να αναπτυχθεί το δυναμικό για την χρηστή διακυβέρνηση και την αηφόρο ανάπτυξη επιτόπου όχι με ένα εμπάγκο αλλά με ένα αηφόρο δράση. Και γνωρίζω ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου η πολιτική επικοινωνία επιβάλλει πολλές φορές υπεραπλούστευση μηνυμάτων όμως θα ενθάρρυνα τους εμπλεκόμενους και τους ευρωβουλευτές. Ίσως να προσπαθούσαμε αυτό το δίλημα της επιλογής μεταξύ εθελοντικού, εθελούσου χαρακτήρα και υποχρεωτικού χαρακτήρα να, να πούμε ότι δεν είναι αυτό το πραγματικό ε, δίλημα. Το δίλημα είναι αποτελεσματική ρύθμιση και κανονισμός και αναποτελεσματική ρύθμιση ή κανονισμός. Αν υπήρχε λοιπόν ε, η δυνατότητα της αποτελεσματικότητας, ε, ο εθελοντικός χαρακτήρας που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διευρυνόμενη η πρόταση αυτή με πολλά άλλα συνοδευτικά μέτρα θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική η προσέγγιση αυτή. Ενώ όπως ακούσαμε η δίσκαμπτη ίσως μόνο υποχρεωτικού χαρακτήρα ρύθμιση μπορεί να μην ήταν εξίσου αποτελεσματική. Θα αποσαφινιστούν αυτά στο μέλλον. Πρόεδρος σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και πάλι για την παρακολούθηση αυτής της ακρόασης και τους ε, επαΐοντες και ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο στην ημερησία διάταξη. Το άρθρο 21 είναι τα διάφορα. Δεν υπάρχουν διάφορα. Και έτσι λοιπόν στις 22 του μήνα που θα είναι η ημερομηνία της επόμενης ε, Συνάντηση 21 και 22 Ιανουαρίου δηλαδή 2015 και εύχομαι με την καινούρια χρονιά να περάσετε πιο πριν υπέροχες χριστουγεννιάτικες διακοπές να χαλαρώσετε και με νέες δυνάμεις να επανέλθετε στο Ευρωκοινοβούλιο την καινούρια χρονιά στην επόμενη συνεδρίαση. Να περάσετε καλά. Γεια σας.